Καλημέρα σε όλους. Να ξεκινήσουμε τις ε, εργασίες μας σήμερα το πρωί. Δυστυχώς κάποιοι από τους προσκεκλημένους μας δεν θα μπορέσουν να έρθουν λόγω της απεργίας ε, που έχει ξεκινήσει από χθες το απόγευμα. Θα ήθελα να ξεκινήσω όμως αμέσως δίνοντας το λόγο στον κύριο Λούντβιξεν ο οποίος είναι εκπρόσωπο. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Λέγομαι Björn Erik Ludvigsen και είμαι νορβηγός αστυνομικός ε, αποσπασμένος στην Interpol. Ήρθα στις αρχές του έτους για να υποστηρίξω το ψήφισμα που έλαβε η Γενική Συνέλευση της Interpol στη Σιγκαπούρη το 2009 που έλεγε, και αυτό ήταν ομόφωνη απόφαση εκ μέρους όλων των χωρών μελών που ήταν παρούσες, ότι οποιαδήποτε μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ε, για την ε, πρόληψη της διανομής ε, παιδικής πορνογραφίας, ακόμα και του μπλοκαρίσματος της πρόσβασης. Γι' αυτό είμαι εδώ, για να σας μιλήσω για αυτό τον κατάλογο domain που διανέμουν πορνογραφικό υλικό με παιδιά στο διαδίκτυο. Πριν ε, μιλήσουμε για την πρόσβαση, θα αναφερθώ σε λίγα τα πιο συγκεκριμένα πράγματα. Το 2004 η Internet Watch Foundation άρχισε να μπλοκάρει παιδικό πορνογραφικό υλικό στο διαδίκτυο. Ε, λίγο αργότερα η νορβηγική αστυνομία ξεκίνησε τα ίδια πράγματα και στα επόμενα χρόνια η Σουηδία, η Δανία, η Φιλανδία και πολλές άλλες χώρες ξεκίνησαν την ίδια διαδικασία. Και μετά ξεκίνησε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα το οποίο λέγεται ΣΕΡΚΑΜ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα ε, κατά της ε, σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών για να προλάβουμε τη διανομή πορνογραφικού υλικού σε όσο το δυνατόν περισσότερες χώρες. Έχουμε 14 χώρες που συμμετέχουν, ε, συμπεριλαμβανομένε και της Europol και της Interpol. Υπάρχει και βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το σύστημα μπλοκαρίσματο ε, βάσει εθνικής νομοθεσίας λειτουργεί σε 8 χώρες αυτή τη στιγμή. Επιπλέον, συνεργαζόμαστε και με χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, ε, όπω για παράδειγμα τη Νέα Ζηλανδία. Αυτό που διαπιστώσαμε στην Ιντερπολ είναι ότι κάποιες χώρες δεν έχουν νομοθεσία που να ορίζει ή να περιορίζει το παιδικό πορνογραφικό υλικό και σε, κάποια νομο... σε κάποιες χώρες ε, δεν αναφέρεται καν στην νομοθεσία. Επομένως ψάχνουμε να βρούμε έναν ελάχιστο κοινό παρανομαστή γι' αυτό που θεωρούμε ότι θα πρέπει να είναι τα λογικά κριτήρια, ε, να γνωρίζουμε όλοι τι είναι η σεξουαλική κακοποίηση και κάναμε ένα κατάλογο αυτών των κριτηρίων που την, ε, τον αποκαλούμε τον κατάλογο των χειρότερων στοιχείων ε, του Ισίντερπολ, που είναι τα ελάχιστα κριτήρια που θα πρέπει να πληρεί κάθε χώρα μέλος για να προστατεύσει ε, τα παιδιά της. Τα παιδιά πρέπει να είναι κάτω των 13 ετών ή να θεωρούνται κάτω των 13 ετών. Στις περισσότερες χώρες ε, ένα παιδί είναι οποιοδήποτε νεότερο κάτω των 18 ετών. Εμείς επιλέξαμε την ηλικία των 13 για να θεωρήσουμε ότι είναι παιδί. Ε, επίσης πρέπει να είναι παιδί, δεν θα πρέπει να είναι σχέδια, άβατερ, ψευδοεικόνες. Ε, πρέπει να φαίνεται ένα παιδί στη φωτογραφία και η φωτογραφία θα πρέπει να είναι ενός πραγματικού παιδιού. Θα πρέπει να υπάρχει σοβαρή κακοποίηση που σημαίνει ε, βιασμός ε, από όλες τις ε, πιθανές ε, διόδους και φυσικά να υπάρχουν και εικόνες. Δεν μιλάμε για φωτογραφίες παιδιών που παίζουν στην παραλία θα πρέπει να υπάρχει διασταύρωση μεταξύ δύο χωρών ή δύο υπηρεσιών, παραδείγματο χάρη τη Δανική Αστυνομία και τη Ιντερπολ, για να αποφεύγονται τα σφάλματα και ε, να είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθούνται τα κριτήρια. Και επίσης πρέπει να υπάρχει διανομή online στο διαδίκτυο παιδικού πορνογραφικού υλικού σε τρεις μήνες και γι' αυτό ε, το όριο των τριών μηνών το επιλέξαμε διότι παρά το γεγονός ότι ορισμένε φορές κάποιοι ιστοσελίδες εξαφανίζονται, διαπιστώνουμε ότι εμφανίζονται σε μια άλλη χώρα ή σε μια άλλη ιστοσελίδα. Γιατί το κάνουμε τώρα αυτό. Αυτό που μπορεί να κάνει η αστυνομία σε οποιαδήποτε εγκληματικό χώρο είναι να προλάβει το έγκλημα. Είναι το πιο φτηνό, έχει τα ελάχιστα δυνατά θύματα και ε, δυστυχώς είναι και το πιο δύσκολο να μετρήσουμε, διότι δεν έχουμε ε, το σενάριο στο οποίο δεν προλάβαμε. Ε, δεν μπορούμε δηλαδή να διαπιστώσουμε κατά πόσο λειτουργεί το σύστημά μας ή όχι. Απλώς κάνουμε εκτιμήσεις. Το κάνουμε για να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των θυμάτων, τα δικαιώματα των θυμάτων που βρίσκονται στις φωτογραφίες, στις ταινίε, μία κακοποίηση η οποία μπορεί να έγινε πριν από κάποιο χρονικό διάστημα, αλλά χρησιμοποιεί χρησιμοποιείται επανειλημμένως και κάποιοι το χρησιμοποιούν για αυνανισμό, για φαντασιώσεις και ορισμένες φορές ε, άτομα τα οποία έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικώς δεν μπορούν να δεχτούν το γεγονός ότι ακόμα και 15 χρόνια μετά κάποιος τους χρησιμοποιεί ως φαντασίωση. Ε, είναι τα παιδιά τους, οι σύζυγοί τους, οι συνεργάτες τους και μπορεί κάποιος να βρει αυτές τις φωτογραφίες στο διαδίκτυο και θέλουμε να προστατεύσουμε και την ιδιωτική του ζωή. Θέλουμε να προστατεύσουμε τη διανομή, και το, <clears throat> τη διανομή του υλικού. Κάθε χώρα που έχει νομοθεσία για το υλικό ε, σεξουαλικής κακοποίησης ε, ε, πρέπει να περιλαμβάνει και κάποια στοιχεία, κυρίως κατάσχεση. Ε, πρέπει να προλάβουμε και την επιζήμια έκθεση στο κοινό. Μπορεί κάποιο να τα δει κατά λάθο γιατί ανοίγουν ε, σελίδε που παίρνουν ε, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή χαζεύουν πορνογραφικό υλικό που μπορεί να, είναι, να ξεκινάει με ενήλικε και μετά να διαπιστώνουν ότι πρόκειται για παιδιά. Ορισμένε φορέ διανέμεται όλο και πιο νέο υλικό και Όλο αυτό φυσικά ε, είναι επιζήμιο για τη ζωή των παιδιών και προσπαθούμε το υλικό αυτό να μην είναι προσβάσιμο ή να μην είναι διαθέσιμο για τους χρήστες. Μας ενδιαφέρει επίσης πάρα πολύ και το χρονικό όριο. Αυτή τη στιγμή έχουμε ε, δισεκατομμύρια χρήστες και ανά δευτερόλεπτο υπάρχει κάτι διαθέσιμο στο διαδίκτυο και μπορούμε ε, να βρούμε ανα πάσα στιγμή τα 2 δισεκατομμύρια ανθρώπους που χρησιμοποιούμε το διαδίκτυο. Ε, το μπλοκάρισμα είναι το πιο ε, ε, αποτελεσματικό. Η διαγραφή είναι χρονοβόρα. Αν γίνει στη χώρα σας και ξέρουμε ποιος ε, φιλοξενεί την ιστοσελίδα είναι πολύ εύκολο. Αρκεί ένα τηλεφώνημα και εξαφανίζεται. Αλλά αν βρίσκεται σε μια χώρα που η πρόσβαση είναι δύσκολη και υπάρχει κάποια διεθνής εγκληματική οργάνωση, δεν έχουν αυτές τις πληροφορίες και φυσικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να διαγραφούν όλα αυτά από το διαδίκτυο. Και όπως σας είπα, κάθε δευτερόλεπτο που είναι διαθέσιμο υλικό στο διαδίκτυο εξακολουθεί να είναι παραβίαση των δικαιωμάτων και της προσωπικής ζωής του ανθρώπου ο οποίος βρίσκεται στις εικόνες της φωτογραφίες. Ε, το πρόβλημα είναι ότι είναι πολύ εύκολο να το μοιραστεί κανείς αυτό το υλικό, να το αντιγράψει, να το αναρτήσει στο διαδίκτυο και αυτό που διαπιστώνουμε είναι ότι αν διαγράψουμε τις φωτογραφίες μέσα σε λεπτά, ώρες ή κάποιες μέρες εμφανίζονται κάπου αλλού, διότι δεν είναι φυσικό μέσο, έχουν εκατοντάδες αντίγραφα και σε κάποιες περιπτώσεις ε, γίνεται και μεταφορά αυτομάτως μεταξύ διαφόρων χωρών για να μην μπορούν ακριβώς να τους εντομήσουν ε, η, η αστυνομία. Εμείς όμως θέλουμε να προστατεύουμε τα θύματα. Ξέρουμε ότι δεν μπορούμε να το καταφέρουμε τόσο εύκολα. Η διαγραφή είναι πάρα πολύ δύσκολη. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε και άλλα μέσα όσο περιμένουμε να γίνει πραγματική ουσιαστική ε, διαγραφή η πρόσβαση δεν βασίζεται σε όρους αναζήτησης. Οποιαδήποτε ιστότοπος βρίσκεται σε κατάλογο έχει ελεγχθεί προσωπικά να δούμε κατά πόσον υπάρχουν τα κριτήρια ή υπάρχει νομοθεσία που να το καλύπτει. Ε, η αστυνομία δεν το κάνει αντί της αστυνόμευσης, θα πρέπει να το κάνει επιπλέον της έρευνας των συλλήψεων, της έρευνας σε σπίτια, κατάσχεση υπολογιστών κλπ. Ξέρουμε ότι δεν είναι η απόλυτη λύση, είναι ένα τμήμα της λύσης. Η πρόληψη είναι τμήμα της λύσης, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να παρεμβαίνουμε και όλα σε κάποιες περιπτώσεις. Όπως πιστεύουν κάποιοι ότι αν μπορεί να το προλάβει δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Αυτό είναι κατάφορο ψεύδος, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να προλάβουμε την κατάσταση. δεν μειώνει το ποσοστό του παιδικού πορνογραφικού υλικού που είναι διαθέσιμο σήμερα στο διαδίκτυο, αλλά μειώνει το ποσοστό του παιδικού πορνογραφικού υλικού που είναι διαθέσιμο για σας σήμερα. Ε, και αυτό είναι το θέμα, ότι δεν μπορεί κάποιος να το βρει, να το φτάσει. Και αυτός είναι ο στόχος μας. Ε, παιδιά τα οποία έχουν αντιμετωπιστεί ε, Ορισμένες φορές προσπαθούμε να βρούμε μία λύση για να τα αντιμετωπίσουμε. Έχουμε αστυνομικού με ε, μικρόφωνα που προσπαθούν ε, να κάνουν μια έρευνα. Εάν μειώσουμε όμως τις έρευνες αυτής της φύσεως θα μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε περισσότερο προσωπικό για να μπορέσουμε ε, να βρούμε τους κακούς, να τους κλείσουμε στη φυλακή και να προστατεύσουμε τα παιδιά μας δεν λειτουργεί με διαφορετικά πρωτόκολλα, δεν, διαφορά με, δεν λειτουργεί με ανταλλαγή υλικού peer-to-peer, -peer, αλλά αλλα κάτι το οποίο μπορούμε να κάνουμε στο διαδίκτυο. Είναι η πιο εύκολη πρόσβαση στο διαδίκτυο. Ε, για τα άλλα πρωτόκολλα θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε άλλα αστυνομικά μέσα. Δεν κάνουμε συλλήψει, δεν μπαίνει κανεί ε, στη φυλακή, δεν ξεκινά καμία αστυνομική υπόθεση. Ε, απλώς προσπαθούμε να ε, κάνουμε πιο δύσκολη την πρόσβαση και έτσι εξοικονομούμε και πόρους διότι θα έχουμε λιγότερες, λιγότερες ιστοσελίδες και την επόμενη φορά που θα κάνουμε μια αντίστοιχη δουλειά. Το μπλοκάρισμα της πρόσβασης δυσκολεύει και τη ζωή των ανθρώπων που ψάχνουν αυτές τις σελίδες. αυτός που έχει το όνομα της σελίδας, ο δικαιούχος της σελίδας είναι υπεύθυνο για αυτό που αναρτάτε. Αν έχετε ένα domain είστε υπεύθυνο για το ε, ε, υλικό που αναρτάτε στο domain σας όπως γίνεται και με μια εφημερίδα. Ε, και προσπαθούμε να εξοικειώσουμε και το κοινό με αυτά τα πράγματα διότι όταν σε κάποιον ε, ε, κόβουμε μία σελίδα έχουμε και μία σελίδα που λέμε ότι τι συνέβη, πότε συνέβη, πού μπορούμε να διαμαρτυρηθούμε αν έχετε domain name τότε μπορείτε να πείτε ότι τι ακριβώς συνέβη. Μπορείτε να διαβάσετε την νομοθεσία της χώρας σα, τα δικαιώματα του παιδιού. Όλοι αυτοί οι σύνδεσμοι που δίνονται, δίνονται αυτές οι πληροφορίε και μπορούν κάποιοι να μάθουν περισσότερο για αυτά τα πράγματα αν θέλουν. It does make it possible by having access blocking. It does it possible for Ορισμένες φορές ε, ε, οι providers μπορεί να αναλάβουν και την ευθύνη από δεντολογική σκοπιά και πολλοί από αυτούς ε, θα σας εκπλήξει αλλά δεν θέλουν να συμμετέχουν στην ε, διανομή πορνογραφικού υλικού στο ε, διαδίκτυο από πλευρά του, ε, αλλά δεν έχουν τρόπο να το προλάβουν. Και ορισμένε φορέ ε, του αρέσει αυτό που κάνει η αστυνομία. Υπάρχουν βέβαια και αυτοί που του αρέσει αυτό που γίνεται και θέλουν να χρησιμοποιούν παιδικό περνογραφικό υλικό. Πολλέ φορέ δεν αρέσει στον κόσμο η αστυνομική μέθοδο. Μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε μια συζήτηση από αυτού. Η μέθοδο αυτή βέβαια επαναξιολογείται συνεχώ κάθε μέτρο επαναξιολογείται. Εμείς αν βάλετε φωτογραφίες ενός 18χρονου και φωτογραφίες ενός 9χρονου που βιάζεται, τότε θεωρούμε ότι αυτό είναι παράνομο και θα μπορέσετε να αναρτήσετε φωτογραφίες κάποιου που είναι ενήλικας και ε, είναι ένα βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου μόνο εάν αφαιρέσετε τη φωτογραφία του 9χρονου. Επίσης δεν θα πρέπει να δεχτείτε σε καμία περίπτωση να υπάρχουν φωτογραφίες ε, και σκεφτείτε να ήταν ένα κατάστημα που να είχε φωτογραφίες ενός παιδιού που βιάζεται. Ακριβώς το ίδιο πράγμα προσπαθούμε να κάνουμε και στο διαδίκτυο. Ως κοινωνία, ως πολιτικοί, ως άνθρωποι δεν δεχόμαστε τη διανομή σεξουαλικού πορνογραφικού υλικού στο διαδίκτυο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Thank you very much. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για την ε, παρέμβαση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Όπως είπαμε ήδη εχθές, ε, θα θέλαμε να σας ζητήσουμε να μας στείλετε τις παρεμβάσεις σας και τις πληροφορίες σας ε, κατά τρόπο ώστε να μπορούμε να ετοιμάσουμε, να εκπονήσουμε ένα κείμενο, θέλουμε να είναι πλήρε και να περιλαμβάνει και τη δική σα συνεισφορά. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Κρίστιαν Χόπ, που εκπροσωπεί mm. την ε, γερμανική αστυνομία. Ζητώ συγγνώμη, θα πρέπει να λείψω για περίπου 20 λεπτά αλλά πρέπει να πάω να ψηφίσω σε μια άλλη επιτροπή. Ανωτέρα βία λοιπόν, θα λείψω για λίγο. Παρακαλώ κύριε Χόπε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Εγώ ε, εκπροσωπώ τι διοκτικέ αρχές της ε, Γερμανίας ε, που ασχολούνται με την έβρεση των ατόμων που κατεβάζουν προγραφικό υλικό θα ήθελα να σας αναφέρω κάποια πράγματα και εγώ για τα domains για να είναι τα πράγματα σαφή. Η, ε, η παιδική πορνογραφία είναι η απεικόνηση της ε, σεξουαλικής εκμετάλλευσης των παιδιών. Όλα όσα βλέπετε στις εικόνες είναι πραγματικότητα. Έχουν συμβεί, έχουν καταγραφεί σε εικόνες η κακοποίηση των παιδιών. Η διαθεσιμότητα και η διάδοση αυτών των εικόνων μέσω του ίντερνετ με εικόνε βία έναντι παιδιών να θυματοποιεί τα παιδιά. Όποιο βλέπει αυτέ τι εικόνε, δηλαδή όταν κάνει κανεί κλικ πάνω στην εικόνα, αποτελεί νέο αδίκημα έναντι αυτού του παιδιού που είναι θύμα. Και αυτό οδηγεί σε μεγαλύτερη ζήτηση. Όσο, όσο περισσότερο κάνει κλικ κάποιο σε μια εικόνα, τόσο περισσότερο παράγεται και τόσο περισσότερο αυξάνονται οι πιθανότητες να υπάρξει περαιτέρω κακοποίηση. Όταν, όταν ανταλλάσσονται αυτές οι εικόνες, επίσης αυτό αποτελεί ε, αδίκημα. Η πλειοψηφία του πορνογραφικού υλικού που αφορά παιδιά παρέχεται μέσω ε, μέσα από διάφορες ε, πηγές στο ίντερνετ. Ανταλλάσσονται οι εικόνες αυτές και όσοι, όσοι, όσοι έχουν, είναι σε θέση να έχουν την ε, δυνατότητα να ε, παράγουν εικόνες μπορούν και να τις ε, λαμβάνουν. Γίνεται λοιπόν αυτή η ανταλλαγή μέσω peer-to-peer -peer to peer ομαδων και η οποιαδήποτε δήλωση αφορά το ποιε είναι οι σελίδες που έχουν τις περισσότερες τέτοιες εικόνες ε, βέβαια δεν νομίζω ότι μπορούμε να το ορίσουμε τελικά αυτό το συγκεκριμένα δηλαδή θέλουμε, τι θέλουμε να μετρήσουμε ακριβώς θέλουμε να δούμε πόσες εικόνες φορτώθηκαν στο ίντερνετ πόσες κατέβηκαν από το ίντερνετ πόσες, ε, πόσα παιδιά είναι θύματα πόσοι είναι οι δράστες είναι πολλά τα ερωτήματα γιατί μιλούμε για διάφορες υπηρεσίες του ίντερνετ που κατέχουν τέτοιο υλικό από το 2000 ε, μιλούμε για εμπορευματοποίηση της, ε, της παιδικής πορνογραφίας. Ε, βεβαίως αυτό μπορεί να διαπιστωθεί μόνο με ότι γίνεται μέσω του ίντερνετ. Το υλικό αυτό συνήθως ανταλλάσσεται δωρεάν. Εκ μέρους λοιπόν των διοκτικών αρχών πρέπει να πω ότι ε, έχουμε τρεις προσεγγίσεις ε, που προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Καταρχήν, πρώτη θέση είναι να ε, βρούμε αυτούς τους δράστες που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης και η αναγνώριση μπορεί να γίνει είτε μέσω του θύματος, αλλά κυρίως ψάχνουμε, και τους, ε, ψάχνουμε τους ίδιους τους ε, δράστες και τις συνθήκες του, ε, κάτω από τις οποίες έγινε το έγκλημα. Προσπαθούμε να αποφύγουμε, να αποτρέψουμε την ανταλλαγή και την παραγωγή τέτοιου υλικού. Επίσης, από, μέσα από έρευνες μπορούμε να ενισχύσουμε την αποτρεπτική δράση άλλων ενδυνάμει δραστών. Προσπαθούμε λοιπόν να δημιουργήσουμε μία σύνδεση ε, μεταξύ και της πρόληψης αλλά και της ε, ε, αύξησης των, τιμών, των ποινών συγγνώμη, ανάλογα με το αδίκημα. Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε την αποτρεπτική διάσταση των δράσεών μας. Σε σχέση και με την αναγνώριση των θυμάτων και των δραστών, έχουμε και το φαινόμενο του grooming, που είναι πολύ σημαντικό η δημιουργία δηλαδή κοινωνικών επαφών μέσω του ίντερνετ, ώστε αυτές να χρησιμοποιηθούν για, ε, για σεξουαλικά εγκλήματα. Αυτό ε, προς το παρόν παραμένει ατιμόρυτο και στη Γερμανία αλλά και ε, διεθνώς και νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να παίξει με καλύτερο ρόλο η αστυνομία. Οι αποδείξεις και οι προθέσεις της ε, σεξουαλικής ε, κακοποίησης ε, είναι πολύ δύσκολο να αποδειχτούν τις περισσότερες φορές. Δεύτερη προτεραιότητά μας για την παιδική πορνογραφία έχει να κάνει με, την, με τους κατόχους και όσους διανέμουν αυτό το υλικό. Όλες οι υπηρεσίες του ίντερνετ μπλέκονται σε αυτό και το Παγκόσμιο Δίκτυο και άλλοι φορείς παροχής τέτοιου υλικού. Ήδη από το 1993 έχουμε ποινικοποιήσει εμείς τέτοια, τέτοιες πράξεις κατοχής υλικού προγραφικού, ε, εικόνων που αποθηκεύονται, βίντεο που αποθηκεύονται στα κομπιούτερ των δραστών. Αυτά αποτελούν ε, αδικήματα. Προσπαθούμε λοιπόν να ενισχύσουμε και τις τεχνικές προδιαγραφές και να δώσουμε νέα, ε, νέους τρόπους λειτουργίας αλλά προσπαθούμε να ε, ενισχύσουμε το ότι πρέπει να περικοποιείται και η κατοχή αλλά και η διανομή συνδέσμων που οδηγούν σε τέτοιες ε, σελίδες πορνογραφικού υλικού. Όταν ε, καθορίζουμε ποιοι είναι οι κάτοχοι και οι διανομής, προσπαθούμε να δούμε ποια είναι τα ίχνη που αφήνουν πίσω τους αυτοί οι δράστες. Προσπαθούμε λοιπόν να έχουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορη ε, ε, έβρεση όλων αυτών των ε, δραστών. Αν όντω καταφέρουμε να βρούμε έναν άνθρωπο που όντω αποδεδειγμένα είναι κάτοχο ή διανομέα τέτοιου υλικού, αυτό έχει μεγάλη σημασία για την περαιτέρω δίωξή του. Τα δεδομένα που έχουμε από, από το ίντερνετ Συνήθω ε, είναι δύσκολο να αναχθούν σε κάποιον συγκεκριμένο ε, κάτοχο, γι' αυτό είναι και δύσκολο για τις ε, διοικητικές αρχές να τον τιμωρήσουν. Ξέρετε ότι στο ίντερνετ υπάρχουν πάρα πολλές κοινότητες γερμανόφωνων, με 300-400 μέλη που δημιουργούνται ακριβώς για να ανταλλάξουν εμπειρίες από σεξουαλικά εγκλήματα. Ε, χωρίς μικρόφωνο ο μιλητής. Diese Boards sind in der Regel sehr abgeschlossen. Man bekommt nur mit Passwort da rein oder mit einer entsprechenden Registrierung. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε κατά πόσο μπορούμε να ε, απελευθερώσουμε τα ε, domains των ε, κατόχων ώστε να μπορέσουμε να βρούμε πού ακριβώς κρύβονται και ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι να τους αναγνωρίζουμε. γρήγορα. Επίσης ε, προσπαθούμε να ε, ποινικοποιήσουμε και την ε, έμεση ή άμεση χρήση και κατοχή τέτοιου υλικού. Το να καταστήσουμε πιο δύσκολη την πρόσβαση σε τέτοιε ιστοσελίδες είναι επίση πολύ σημαντικό και υπάρχει στη Γερμανία αυτή τη στιγμή και συγκεκριμένη νομοθεσία Βεβαίως αυτό έχει να κάνει και με την ε, διατάραξη της ε, δημοσίας ε, ασφάλειας. Προσπαθούμε λοιπόν να συνδέσουμε όλα αυτά τα αδικήματα και να ενισχύσουμε και τις αστυνομικές αρχές οι οποίες πρέπει να μπορούν να παρεμβαίνουν και να αναλαμβάνουν αποτρεπτικά μέτρα για τους κατόχους του πορνογραφικού υλικού. προσπαθούμε να δυσκολέψουμε την ε, επαφή ε, των δραστών με τα θύματα. Ε, προσπαθούμε να αποτρέψουμε την θυματοποίηση των παιδιών. Και βεβαίως αυτό έχει να κάνει με το ότι αν ένα παιδί ε, έχει, τύχει, έχει πέσει θύμα ε, σεξουαλικής κακοποίησης ε, και μεγαλώσει κάποια στιγμή μπορεί να βρεθεί αντιμέτωπο με τις δικές του εικόνες από τότε που ήταν παιδί και να δημιουργηθούν σημαντικά ψυχολογικά προβλήματα. Προσπαθούμε λοιπόν να δυσκολέψουμε την επαφή των ανθρώπων αυτών με τα θύματα για να μην τα τραυματίζουν. Μέσα σε τέσσερις εβδομάδες είδαμε ότι υπήρξε μία ιστοσελίδα η οποία είχε 1.250.000 επισκέψεις μέσα σε τέσσερις εβδομάδες. Αυτό λοιπόν είναι σημαντικό δεδομένο, το οποίο φυσικά αποτελεί αδίκημα και επισύρει βαριές ποινές. Ο νόμος που έχουμε θεσπίσει στην Γερμανία ισχύει με ένα ιδιαίτερο τρόπο γιατί και αφορά την διαγραφή των ιστοσελίδων. Οι ιδιωτικές αρχές ήδη έχουν ε, καταγεγραμμένες τις ιστοσελίδες που μας έχουν ε, ανακοινωθεί και έχουμε διαγράψει τις ιστοσελίδες που περιείχαν πορνογραφικό υλικό. Προσπαθήσαμε να διακόψουμε την παροχή αυτού του υλικού και μέσω των γνωστών διόδων που υπάρχουν, προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε και με τις εθνικές αρχές της των ΗΠΑ και με τη Ρωσία, με τις ε, επίσης ε, αρμόδιες αρχές που βρίσκονται εκεί. Στην, ε, η, δυσκολία, λοιπόν στην πρόσβαση αποτελεί μια συμπλήρωση, όχι εναλλακτική στη διαγραφή η δυσκολία πρόσβασης θα πρέπει να ισχύει μέχρι να φτάσουμε στο σημείο της διαγραφής αυτής της ιστοσελίδας. Η διαγραφή είναι το, η πρώτη μας επιλογή και η δυνατότητα, η διακοπή της πρόσβασης είναι η παραπληρωματική ενέργεια που έχουμε λάβει. Επίσης πρέπει να δούμε ποιο είναι το χρονικό περιθώριο που μπορούν ε, να είναι διαθέσιμες αυτές οι ιστοσελίδες ε, από τη στιγμή που καταγράφονται ως ε, σελίδες πορνογραφικού υλικού ώστε να μπορεί να παρέμβει η αστυνομία. Προς το παρόν, κάθε μήνα έχουμε περίπου 160 αναφορές για πορνογραφικές σελίδες με υλικό, με εικόνες από παιδιά. Ε, οπότε τώρα το ερώτημα είναι αν αυτές οι 160 σελίδες μπορούν να διαγραφούν μέσα σε 24 ώρες. Περίπου 40% μετά από 7 ημέρες βρίσκονται διαθέσιμοι στο ίντερνετ. Διαγράφονται και μετά από 7 μέρες επανεμφανίζονται στο ίντερνετ και οι δράστες μπορούν να τις ε, ξαναεπισκεφθούν. Με βάση λοιπόν όλα αυτά, από τη, έτσι όπως το βλέπει η αστυνομία και οι διοκτικές αρχές, ε, η ε, προσπάθεια ε, του να δυσκολεύσουμε την πρόσβαση στις ελευθεραπτές, αυτές είναι ένα αρκετά σημαντικό εργαλείο που έχουμε. Αν, ε, παρόλο που επιτυγχάνουμε μόνο την ε, διαγραφή ενός μικρού τμήματος των ιστοσελίδων αυτών, παρόλα αυτά αυτές περιλαμβάνουν ένα πολύ σημαντικό αριθμό φωτογραφιών και γενικώ υλικού. Οπότε είναι σημαντική η προσπάθεια που γίνεται. Ένα παρόμοιο εργαλείο είχαμε και με τις κλοπές οχημάτων. Φυσικά η, η παιδική πορνογραφία είναι παγκόσμιο φαινόμενο. Προσπαθούμε με, το, με τα εργαλεία που έχουμε και με διεθνή συνεργασία να το αντιμετωπίσουμε και προσπαθούμε να έχουμε δικτύωση με τις διάφορες εθνικές αρχές. Φυσικά είναι ιδιαίτερο το θέμα αυτό και δεν πρέπει να ξεχνούμε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του η βιομηχανία νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει ακόμη περισσότερο με την τεχνογνωσία της και με τις υπηρεσίες της. Ας πούμε οι providers του ίντερνετ μπορούν να βοηθήσουν. Γιατί υπάρχουν πολλές καλές προσεγγίσεις ε, και με τις γραμμές βοηθείας έχουμε δει πολύ καλά αποτελέσματα και σε αυτά προσπαθούμε να βασιστούμε. Ευχαριστώ. Ε, ε, Ευχαριστώ για την παρουσίασή σας. Να δώσουμε τώρα το λόγο στην κυρία Σό. Good morning. Καλημέρα. Λέγομαι Γαβριέλα Σό από την Μονάδα Προστασίας Παιδών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το κέντρο αυτό είναι μια ειδική υπηρεσία των διοκτικών υπηρεσιών και των σωμάτων ασφαλείας για να καταπολεμήσει την σεξουαλική κατάχρηση και εκμετάλλευση παιδών. Λόγω του ότι διαπιστώσαμε αυξημένες τέτοιες περιπτώσεις μέσω του ίντερνετ και επιζητούμε επίσης να καταπολεμήσουμε και την εκμετάλλευση παιδών στο ίντερνετ. Είναι δηλαδή ένα κεντρικό σημείο συνεννόησης και ανταλλαγής πληροφοριών. Απλοί πολίτες μπορούν με ένα, μέσω του διαδικτύου με ένα απλό κομβίο που μπορούν να πιέσουν στην ιστοσελίδα μας να καταθέσουν πληροφορίες για τοποθεσίες που, όπου εμφανίζεται παιδική πορνογραφία αλλά και άλλες μη κυβερνητικέ οργανώσεις και ακόμη και αστυνομικές υπηρεσίες μας υποβάλλουν στοιχεία. Δεχόμαστε χιλιάδες αναφορές κάθε χρόνο που αφορούν ιδιαίτερα ε, κλήσεις μέσω του ίντερνετ για την εκμετάλλευση παιδών. Επίσης είμαστε ιδρυτικό μέλος της Global Task Force που είναι μία οργάνωση που συγκεντρώνει τέτοια στοιχεία διεθνώς και τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουμε γίνει ειδικευμένη διοκτική υπηρεσία εμπειρογνώμων για τέτοιες περιπτώσεις παιδικής εκμετάλλευσης. Επίσης συμμετέχουμε σε χρηματοδότηση από την Κομισιόν σε ένα πρόγραμμα που μόλις συμπλήρωσε την πρώτη του πειραματική φάση. Και εμείς δεχόμαστε το σχέδιο οδηγίας που συζητάτε ή τα, τα μέτρα που προτείνετε μάλλον για την καταπολέμηση της εκμετάλλευσης των παιδιών. Γιατί νομίζουμε ότι θα επιτρέψει την επιτυχή καταπολέμηση τέτοιων πρακτικών και θα διευκολύνει την καταδίκη και δίωξη των υπευθύνων. Πρέπει να γνωρίζουμε βέβαια ότι δεν είναι ουδέτερος χώρος το ίντερνετ. Υπάρχει ένα ιδιαίτερο τμήμα του που αφορά ακριβώς τα παιδιά και η ανωνυμία του κυβερνοχώρου καθιστά τα παιδιά ιδιαίτερα ευάλωτα σε εκμετάλλευση. Γι' αυτό δεχόμαστε και το άρθρο 6 για τις προσκλήσεις παιδών σε σεξουαλική χρήση και εκμετάλλευση. Το λεγόμενο grooming που οδηγεί τα παιδιά προς σεξουαλικές επαφές είτε μέσω είτε έξω του διαδικτύου προσπαθώντας να μειώσει τα αισθήματα εδούς τους για να τα καταστήσει χρήσιμα στον εκμεταλλευτή. Δημιουργείται λοιπόν ένα περιβάλλον συζήτησης online ώσπου να πιστεί το παιδί. Πρέπει βέβαια να γνωρίζουμε ότι σε μερικές περιπτώσεις, πολλές μάλιστα, το θύμα δεν οθείται προς μια συνάντηση εκτός ίντερνετ αλλά μέσω μιας απλής webcam. Είναι απαράδεκτο να υπάρχει τέτοια διαδραστικότητα στο διαδίκτυο για σεξουαλική κατάχρηση των παιδιών. Επίσης το άρθρο 10 δεχόμαστε για τις απαγορεύσεις περαιτέρω χρήσης σελίδων όσων έχουν καταδικαστεί για τέτοια πρακτική. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε αυτούς πρόσβαση καν σε ιστοσελίδες με παιδιά ή σε παιδιά γενικότερα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο όσοι έχουν καταδικαστεί για σεξουαλική κατάχρηση παιδών εγγράφονται σε ένα ειδικό μητρό για να μπορεί να παρεμποδιστεί νομικά η σχέση τους με παιδιά. Πρώτο καθήκον βέβαια είναι να τους ταυτίσουμε και να τους απαγορεύσουμε τη χρήση επαγγελμάτων που αφορούν παιδιά. 60.000 ενήλικες σε τρία χρόνια από το μέχρι το 2007 έχουν έτσι παρεμποδιστεί νομικά από εργασία που αφορά παιδιά, που έχει σχέση με παιδιά. αυτοί είχαν προσπαθήσει εσκεμένα να βρουν μια θέση εργασίας που να αφορά παιδιά. Αυτά όλα πρέπει να απαγορεύονται. Οποιαδήποτε δυνατότητα επαφής με παιδιά επαγγελματικά. Έχει δημιουργηθεί μια ειδική ομάδα σε συνεργασία με άλλες υπηρεσίες του Ηνωμένου Βασιλείου που συμπεριλαμβάνει και την καταπολέμηση της αδείας εξόδου πολιτών που βγαίνουν από το Ηνωμένο Βασίλειο για δεδηλωμένους σκοπούς σεξουαλικής εκμετάλλευσης. Έτσι ελπίζουμε όσοι ταξιδεύουν σε άλλες χώρες για να έχουν πρόσβαση σε σεξουαλικά σε παιδιά να μπορούν να παρεμποδιστούν οι μετακινήσεις αυτές. Με τέτοια μέτρα νομίζουμε ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Επίσης το άρθρο 21 για το μπλοκάρισμα της πρόσβασης σε ιστοσελίδες που επιδεικνύουν σεξουαλική χρήση παιδιών. Είναι κάτι που το δεχόμαστε. Α, θα πρέπει να συζητηθεί περαιτέρω ο ακριβής τρόπος. Ορισμένοι που επικρίνουν το άρθρο 21 λένε ότι το μπλοκάρισμα δεν είναι αποτελεσματικό εφόσον αλλάζουν οι εικόνες από σελίδα σε σελίδα. Εμείς θα θέλαμε να τονίσουμε ότι η διανομή τέτοιων φωτογρα... πορνογραφικών φωτογραφιών με παιδιά με βάση την τεχνολογία peer-to-peer -peer, είναι κάτι που πρέπει και μπορεί να απαγορευτεί γιατί αυτά τα δίκτυα λειτουργούν μέσω της συνεννόησης ανθρώπων που έχουν την ίδια νοοτροπία και η παραγωγή νέων φωτογραφιών μέσα των δικτύων αυτών peer-to-peer -peer to peer μπορει να παρακολουθηθεί με επιτυχία. Γι' αυτό ζητούμε από τις χώρες μέλη να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους να συρθούν στη δικαιοσύνη όσοι εκμεταλλεύονται παιδιά και μέσω της τεχνολογίας peer-to-peer. -peer. to peer αυτά το μπλοκάρισμα πρέπει να τονίσουμε ότι είναι μία αποτελεσματική μέθοδος. Γιατί αν γνωρίζουν όσοι έχουν καταδικαστεί ότι θα φανεί η πρόσβασή τους και μέσω peer-to-peer σε τέτοιες ιστοσελίδες θα, υπα... αυτό... θα αποτελέσει αυτό ένα αποτελεσματικό αντικίνητρο. Θα ξέρουν δηλαδή ότι μπορεί να αναγνωριστεί η δραστηριότητά τους αυτή και να γίνει γνωστή. Το είπαν και άλλοι ομιλητές ότι το μπλοκάρισμα της πρόσβασης εμποδίζει την περαιτέρω εκμετάλλευση παιδιών που έχουν ήδη τύχη τέτοιας Η καταστροφή τέτοιων ιστοσελίδων είναι κάτι που μπορεί να επιδευτεί και πολύ σύντομα μάλιστα. Αυτό είναι προτιμότερο από την, το μπλοκάρισμα της πρόσβασης, αλλά που μπορεί να παραμείνει μια τακτική τουλάχιστον χρήσιμη. Βραχυπρόθεσμα. Ευχαριστώ. Και εμείς σας ευχαριστούμε κυρία Σόουλ. Τώρα θα δώσω το λόγο στην κυρία Μπάιλα. Καλημέρα. Είμαι ψυχολόγος πολλά χρόνια και εργάζομαι με παιδιά που έχουν κακοποιηθεί σεξουαλικώς εδώ και 20 χρόνια περίπου. Και νομίζω ότι αυτό που λείπει από τη συζήτηση είναι ε, η άποψη του θύματος. Εγώ λοιπόν θα αλλάξω λίγο την ομιλία που είχα ετοιμάσει και θα προσπαθήσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς συζητάμε και έτσι μπορεί να απαντήσω και κάποια από τα ερωτηματικά που ετέθησαν εχθές. Έστω ότι έχουμε ένα μικρό κοριτσάκι, ένα μικρό αγοράκι, 6 χρονών, πηγαίνει δημοτικό σχολείο, πήγε στον επιαγωγείο και εκεί έκανε ένα μάθημα όπου ή το αγοράκι το κοριτσάκι έμαθε να λέει όχι εάν κάποιος προσπαθήσει να τους αγγίξει με τρόπο που δεν επιτρέπεται. Πηγαίνει στο δημοτικό σχολείο, ε, οι γονείς του δουλεύουν και έχουν αυτό τον καταπληκτικό φίλο στη γειτονιά, τον οποίο ας ονομάσουμε Τζον. Οι γονείς είναι ανακουφισμένοι διότι ο Τζον προσφέρεται να κάνει babysitting, ε, φροντίζει και λίγα πράγματα στο σπίτι και είναι πάρα πολύ χαρούμενοι γιατί φροντίζει πραγματικά το παιδί τους. Και Κάποια στιγμή αρχίζει να αγγίζει το παιδί και το παιδί έχει πρόβλημα διότι υπάρχει αυτός ο καταπληκτικός τύπος που τον γνωρίζει, ξέρει ότι οι γονείς μου το συμπαθούν και σε ποιον θα το πω. Ακόμα και αν το πω στη μαμά μου, δεν θέλω, ε, ότι δεν θέλω να το κάνει αυτό, δεν μπορεί να φανταστεί πόσο ντρέπομαι μαμά μου. Έτσι ο Τζον συνεχίζει και κακοποιεί το αγοράκι ή το κοριτσάκι. το κακοποιεί στοματικά, προκτικά και φυσικά ε, δεν ε, μπορεί να σταματήσει να κάνει πράγματα και του αρέσει ε, ο Τζον ως άνθρωπος αλλά δεν του αρέσει αυτά που κάνει. Θέλει απλώς ο Τζον να σταματήσει να κάνει αυτά που κάνει όταν το πονάει. Αλλά αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πει. Τα παιδιά λοιπόν δίνουν κάποιες ε, ενδείξεις ε, ώστε να καταλάβει κάποιος τι συμβαίνει αλλά κανένας δεν μπορεί να το κατανοήσει, δεν μπορεί να φανταστεί ότι στη γειτονιά μου, στην οικογένειά μου, στο ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον γνωρίζω κάποιον ο οποίος κακοποιεί παιδιά δούμε τα στατιστικά στοιχεία, πρέπει να παραδεχτούμε ότι κατά πάσα πιθανότητα ακόμα και εδώ στην αίθουσα υπάρχουν και θύματα, αλλά ίσω και δράστε οι οποίοι δεν εντοπίστηκαν ποτέ. Και αυτό είναι αυτό που συζητάμε και αυτό είναι αυτό που δεν θέλει κανεί από εμά να δεχτεί. Τελικά, το παιδί συνειδητοποιεί ε, καθώς μεγαλώνει και η κακοποίηση συνεχίζεται ε, και τα παιδιά δυστυχώς αντιγράφουν. Και το μικρό γοράκι, το μικρό κοριτσάκι διαπιστώνει ότι ε, ε, ο Τζον πλέον βγάζει φωτογραφίες ή κάνει ταινίες και τα πράγματα δυσκολεύουν γιατί τώρα το εκβιάζει και του λέει αν το πεις θα τους δείξω και αυτή την ταινία και η ταινία θα τους δείξει ότι το ήθελες και κανένας δεν θα σε πιστέψει ότι δεν ήθελες. Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι αν εμείς ως ενήλικες δεν φροντίζουμε τα παιδιά και αν εμείς ως ενήλικες δεν αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε τι ακριβώς είναι αυτό που συζητάμε και το γεγονός ότι οι άνθρωποι στο ευρύτερο περιβάλλον μας κάνουν αυτό που θέλουν να κάνουν με τα παιδιά γιατί εμείς δεν προσέχουμε αρκετά, δεν θα αλλάξει τίποτα γιατί αυτό το μικρό αγοράκι ή το μικρό κοριτσάκι μπορεί να πει όχι στον Τζον αλλά ε, ο Τζον δεν ακούει. Τα παιδιά λοιπόν χρειάζονται έναν ενήλικα που να τους φροντίζει. Εάν στη συνέχεια οι εικόνε αυτές διανέμονται στο διαδίκτυο ή μέσω δικτύων peer-to-peer, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα για το παιδί, όπως είπαν και οι προλαλήσαντες, διότι πλέον η ντροπή είναι δημόσια. αυτό που είναι το χειρότερο για μένα ε, είναι πλέον δημόσιο και δεν ελέγχω ποιο το βλέπει. Κανένα δεν βλέπει τι μου Βλέπουν όλοι συγγνώμη, τι μου συνέβη όταν ήμουν 6 χρονών. Και για να είμαι ειλικρινή, ακόμα και αν διαγράψουμε αυτέ τι ιστοσελίδε, δεν μπορούμε να είμαστε βέβαιοι ότι δεν θα ξανακυκλοφορήσουν αυτέ οι φωτογραφίε ε, είτε μέσω του διαδικτύου είτε μέσω δικτύων peer-to-peer, γιατί δεν ξέρουμε ποιο έχει τι στον υπολογιστή του και με ποιον το μοιράζεται. Το ίδιο ισχύει και για το grooming. Αν εγώ είμαι ε, στην προεφηβική φάση, είμαι 12 χρονών, έχω προβλήματα με τους γονείς μου, γιατί αυτό είναι η εφηβεία, προβλήματα και για τους γονείς αλλά και για τα παιδιά. Και ε, είναι κάποιο στο διαδίκτυο ο οποίο λέει κάποια ψέματα, αλλά δεν είναι κάτι φρικτό. Μπορεί να είναι 40 και να λέει ότι είναι 30. Μπορεί να είναι παντρεμένο και να έχει τρία παιδιά και να μην το λέει. Αλλά αυτό που κάνει στο διαδίκτυο είναι ακριβώ αυτό που έκανε και ο ε, Τζον όταν ε, ήταν δίπλα μου. Θα ξεκινήσει η σχέση μαζί μου και θα βρεθώ αντιμέτωπο με πράγματα τα οποία δεν θέλω να αντιμετωπίσω. Αλλά δεν ξέρω πώς να το αντιμετωπίσω. Διότι έχω ε, εκπλαγεί, ξέρω ότι πρέπει να το πω στους γονείς μου, αλλά πώς θα το πω στους γονείς μου ή ακόμα και στο δάσκαλό μου ότι υπάρχει αυτός ο τύπος με τον οποίο κάνω τσάτ εδώ και τρεις μήνες που τώρα ε, έχει αρχίσει να μου κάνει σεξουαλικές προτάσεις, με εκβιάζει και μου ζητάει να γδυθώ μπροστά σε ε, ε, κάμερα, να αυνανιστώ μπροστά στην κάμερα και μου λέει μετά ότι αν το πεις αυτό, εγώ θα της δείξω τις φωτογραφίες και κανένας δεν θα πιστέψει ότι δεν το θέλεις. Εγώ έχω πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα και αν ο περίγυρός μου δεν αντιληφθεί ότι δεν φταίω εγώ, γιατί εγώ είμαι 12 χρονών, Ακόμα και αν το πω ε, και είμαι ένα παιδί που είμαι έξυπνο και ε, έχω και το θάρρος τη γνώμη μου, δεν έχω κανένα όπλο ενάντια σε έναν άνθρωπο που με σεξουαλι... Ε, κακοποιεί σεξουαλικά. Δυστυχώ πρέπει να το παραδεχτούμε ότι πάντα, τα πάντα είναι υπέρ του ενήλικα που κακοποιεί τα παιδιά. Και αυτό το οποίο δεν αντιλαμβανόμαστε είναι σεξουαλική κακοποίηση από γυναίκε. Και υπάρχει, αλλά κανένα δεν θέλει να το συζητήσει. Ε, διότι όλε είναι δυνητικά μητέρε και η κάθε μητέρα είναι δυνητικά καλή μητέρα. Και αυτό είναι μια πτυχή που πρέπει να λάβουμε υπόψη και πρέπει να το γνωρίζουμε διότι είναι κάτι πάρα πάρα πολύ δύσκολο. Το να πούμε ότι χρειαζόμαστε περισσότερη πρόληψη είναι κάτι που με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη. Αλλά η πρόληψη δεν θα έχει κανένα αποτέλεσμα εάν δεν εστιάσουμε στη σωστή διαπαιδαγώγηση και φροντίδα των παιδιών μας. Πρέπει να τα διδάξουμε, πρέπει ως ενήλικες να τους ε, μάθουμε έναν τρόπο σκέψης ώστε να μην... Ε, ε, βρεθούν σε πανικό ή σε ιστερία, αλλά να μπορέσουν να ε, ελέγξουν την κατάσταση όταν προκύψει το πρόβλημα. Διότι πρέπει να είμαστε ειλικρινεί. Εάν μιλάμε για παράδειγμα για τον αδερφό μου, δεν θέλω καν να φανταστώ ότι ο αδερφό μου είναι βιαστή ανηλίκων. Εάν ε, όμω ένα παιδί μου, θε, μου πει ότι δεν θέλω να κάνω παρέα με το θείο του μου, πρέπει να βρω για ποιο λόγο δεν θέλει να κάνει παρέα μαζί. Τι συμβαίνει. Στη Γερμανία είχαμε 11.961 καταγγελίες στην αστυνομία. Αυτό το στοιχείο σημαίνει ότι κάθε μέρα έχουμε 32 παιδιά τα οποία επισήμω κακοποιούνται σεξουαλικώ. και αυτέ είναι μόνο οι περιπτώσει που καταγγέλλονται επισήμω στην αστυνομία. Ελπίζω να μπορέσετε να καταλάβετε γιατί είναι τόσο δύσκολο για τα παιδιά ακόμα και να το αποκαλύψουν και ακόμα πιο δύσκολο να καταλήξει αυτό στην αστυνομία. Τα πραγματικά στοιχεία δεν τα γνωρίζουμε και δεν θα τα μάθουμε ποτέ. Αλλά Εάν δεν αρχίσουμε να αντιδρούμε τώρα και αν δεν αρχίσουμε να εναρμονίζουμε την ομοθεσία μας και δεν αρχίσουμε να ε, ε, ελέγξουμε τα πράγματα που γνωρίζουμε σήμερα χωρίς να λάβουμε τα μέτρα που απαιτούνται ώστε να προστατεύσουμε τα παιδιά μας σήμερα αλλά και στο μέλλον τότε θα πρέπει πραγματικά να ντρεπόμαστε για τους εαυτούς μας. Δεν μπορεί να λέμε ότι τα παιδιά είναι το μέλλον μας γιατί δεν τα φροντίζουμε όπως πρέπει. Υπάρχουν καταπληκτικά παιδιά που ε, θα μιλήσουν, ε, έχουν ένα υπέροχο οικογενειακό περιβάλλον, αλλά υπάρχει και ένα υψηλό ποσοστό παιδιών που δεν έχουν σε ποιον να στραφούν. Και αυτά τα παιδιά θα πρέπει να προσεγγίσουμε, αυτά τα παιδιά είναι αυτά τα οποία θα πρέπει να προσέξουμε λίγο περισσότερο. Γι' αυτό ακριβώς ε, το ε, Innocence in Danger εκτιμά πάρα πολύ την οδηγία. Πιστεύουμε ότι υπάρχουν κάποιε λεπτομέρειε οι οποίε χρήζουν βελτίωση, αλλά αν δεν προχωρήσει αυτή η οδηγία, νομίζω ότι πρέπει να γυρίσουμε σπίτι μα και να πούμε στα παιδιά μα, ξέρει, δεν κάναμε και πολύ καλά τη δουλειά μα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και τώρα Ο κύριος Πιόρν Σέλστρομ, εκπρόσωπος της ε, Σουηδικής Αστυνομίας. Παρακαλώ. Good morning everybody. Καλημέρα σας. Όπως γνωρίζετε λέγομαι Σέλστρομ και είμαι επικεφαλής της ομάδας καταπολέμησης της παιδικής εκμετάλλευσης στη Σουηδία. Χαίρομαι ιδιαίτερα για την παρουσία μου εδώ και για το γεγονός ότι ενδιαφέρεστε και εσείς εδώ κάτω για τα προβλήματά μας στο βορρά εκεί απάνω. Δεν είναι πολλά δέκα λεπτά βέβαια, θα προσπαθήσω όμως να τα σεβαστώ. Τα θα σεβαστώ, θα σεβαστώ. Τι να κάνω. Η Σουηδία έχει πολλές φορές προσπαθήσει να συνεργαστεί και με προμηθευτές πρόσβασης για να μπλοκάρει ιστοσελίδες παιδοπορνογραφίας και έχει εξετάσει 5 με 90% των καταναλωτών και καταναλωτριών. Η δουλειά αυτή είναι απλή και δεν κοστίζει και πολύ. Το μπλοκάρισμα είναι κάτι που γίνεται πολύ εύκολα. Στις αρχές της συνεργασίας μας αυτής τέθηκαν μερικά προβλήματα όπως για την ελευθερία του λόγου και τον αρνητικό χαρακτήρα που θα είχε η λογοκρισία σε εισαγωγικά. Αλλά τελικά πίστηκαν όλοι ότι είναι χρήσιμο αυτό ως μέσο για την καταπολέμηση της παιδοπορνογραφίας. Μας έχουν βρήσει πολλές φορές και με άσκημο τρόπο Αλλά το θέμα είναι ότι εδώ δεν πρόκειται καθόλου για ελευθερία του λόγου, ούτε για λογοκρισία, αλλά για παρεμπόδιση της διάδοσης φωτογραφιών και άλλου υλικού που αφορούν εκμετάλλευση παιδιών. Εγώ δεν καταλαβαίνω πώς μπορούν μερικοί να αρνούνται το μπλοκάρισμα τέτοιων ιστοσελίδων. Δεν νομίζουμε ότι είναι πρόβλημα το μπλοκάρισμα για το ίντερνετ. Και έχω την εντύπωση ότι όσοι μας επικρίνουν έχουν πάψει πια να το πράττουν. Παρ' όλα αυτά, με χαρά θα δεχόμασταν κάποιο τρίτο αουδέτερο ανεξάρτητο οργανισμό να ελέγξει τις δραστηριότητες μας. Επίσης συνεργαζόμαστε με τον χρηματοπιστωτικό τομέα για να παρεμποδίσουμε πληρωμές από και προς εμπορικές παιδοπορνογραφικές ιστοσελίδες. Έχουμε συνεννοηθεί με τις κυριότερες τράπεζες στη Σουηδία και τις κυριότερες πιστωτικές κάρτες. οι εμπορικές ιστοσελίδες που προμηθεύουν τέτοιο υλικό έχουν μειωθεί πολύ αλλά παρόλα αυτά θα μπορούσαμε να εφαρμόσουμε ανα πάσα στιγμή αν ξανααυξηθεί ο ρυθμός τους την ίδια συμμαχία που σας ανέφερα προηγουμένως. Και αυτό η παρεμπόδιση των πληρωμών δηλαδή είναι κάτι που γίνεται πολύ εύκολα και φτηνά. Και αν δεν αρκεί ούτε αυτό Είμαστε και εμείς μέλος της European Financial Coalition για την οποία μίλησε η κυρία Σο και κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ταυτίσουμε και τα παιδιά αυτά που την χάνουν εκμετάλλευσης. Ξέρει κανείς από εσά πόσα από αυτά τα εκατομμύρια παιδιών είναι γνωστά. Είναι κανείς που το ξέρει. 1852 μόνον τέτοιες περιπτώσεις γνωρίζει η Ιντερπόλ. 1852 παιδιά έχουν ταυτιστεί παγκοσμίω μόνο. Αλλά βεβαίως είναι πολύ περισσότερα τα θύματα. Η ταύτιση αντίθετα από όσα είπα προηγουμένως είναι δύσκολη δουλειά και χρειάζεται και διεθνή συνεργασία. Εμείς είμαστε υπέρ της πρωτοβουλίας αυτής του Κοινοβουλίου γιατί θεωρούμε ότι αν οι χώρες μέλη δεν έχουν πια καμία δικαιολογία για να καταπολεμήσουν, για να αναρνηθούν την καταπολέμηση των ιστοσελίδων αυτών, τότε θα διευκολυνθεί και από τους προμηθευτές της πρόσβασης η εφαρμογή της νομοθεσίας και θα σιωπήσουν όλοι όσοι επικρίνουν την καταπολέμηση, αν και στη Σουηδία αυτό δεν συμβαίνει πια. Η νομοθεσία αυτή επίσης θα πείσει ακόμα και τους μικρότερους προμηθευτές που θεωρούν ότι όλα πρέπει να είναι ελεύθερα στο ίντερνετ και ανεξέλεγκτα. Δυστυχώς βέβαια μπορεί μερικοί να ζητήσουν να συνεργαστούμε για την καταπολέμηση και άλλου είδους εγκληματικότητας, αλλά εμείς δεν συμφωνούμε. Πρέπει να παραμείνει ειδικά επικεντρωμένη προσοχή μας σε αυτό το θέμα. Δεν υπάρχει καμία δικαιολόγηση τέτοιων δραστηριοτήτων με επιχειρήματα copyright ας πούμε. Πριν από μερικά χρόνια στο γερμανικό τύπο μου είχα γράψει κάτι ή μάλλον μου είχαν πάρει μια συνέντευξη και είχα πει ότι δυστυχώς ό,τι για να έχουμε πετύχει δεν αρκεί διότι λίγες χώρες μόνο στον κόσμο χρησιμοποιούν την τεχνολογία του μπλοκαρίσματος. Πρέπει περισσότερες χώρες να εφαρμόσουν ανάλογα μέτρα είναι σαν τον πίθο των Δαναίδων. Δεν αρκεί να βουλώσουμε μερικές τρύπες στον πίθο αυτό, αλλά όλες. Θα συνεχίσουμε πάντως τις προσπάθειές μας και θα τις αυξήσουμε για να πάψει η διάδοση τέτοιου υλικού. Αλλιώς δεν χρειάζεται καν να ασχοληθούμε και θα το συνεχίσουμε όχι για το δικό μας και το δικό σας συμφέρον αλλά για τον παιδόν διότι κάλιο αργά παρά ποτέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Νομίζω ότι τώρα μπορούμε να ξεκινήσουμε το δεύτερο τμήμα των εργασιών σήμερα το πρωί, να δώσω το λόγο στην κοινωνία των πολιτών πλέον, στις οργανώσεις που είναι εδώ και των πολιτριών και στις οργανώσεις που είναι εδώ παρούσες σήμερα και από εκεί και πέρα να ακούσουμε ερωτήσεις ε, από τους ευρωβουλευτές. Υπάρχουν ερωτήσεις? Όχι, δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Ο κύριος Μπρόντς, παρακαλώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ο κύριος Χόπερ αναφέρθηκε στους service providers και στους χρήστες. Ε, συγγνώμη, δεν κατάλαβα τι ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η διαφορά που είπατε εκεί, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό που ρωτώ είναι όλοι αυτοί ε, ενσυνείδητα διαβιβάζουν το υλικό αυτό ή κατά λάθο ή μπορεί να είναι και απολύτω αθώοι σε κάποιες περιπτώσεις γιατί δεν, απολύτως, δεν κατάλαβα απολύτως τι εννοούσατε. Η κυρία Σό επίσης μίλησε για καταγεγραμμένους ε, εγκληματίες ε, σεξουαλικών πράξεων που έχουν πρόσβαση σε παιδιά λόγω καταλαβα απολυτω τι επαγγελματός τους. για καταγεγραμμενους εγκληματιε ερώτημα που εχουν προσβαση σε παιδια λογω του επαγγελματό του. ενα ερωτημα που προκυπτει ειναι το εξή. Τι γίνεται με αυτούς τους καταχωρημένους που ψάχνουν να βρουν δουλειά ειδικά ε, κοντά σε παιδιά. Αυτοί έχουν, ε, θεωρούνται εγκληματιές. Και δεύτερον, οι καταγεγραμμένοι αυτοί ε, δεν πρέπει να έχουν ε, να, απαγόρευση πρόσβαση στο ίντερνετ. Υπάρχει κάτι τέτοιο. Επίσης, Ακούστηκε ότι οι εγκληματίες αυτοί είναι συνήθως άνθρωποι εμπιστοσύνη. Και τα παιδιά πιστεύουν ότι δεν θα τα πιστέψουν αν ε, καταγγείλουν κάτι τέτοιο. Ξέρω κι εγώ μια παρόμοια περίπτωση που αυτό ακριβώς συνέβη. Και το παιδί δίκιο είχε ότι δεν θα το πίστευαν. Υπάρχουν ε, περιπτώσεις συζύγων των εγκληματιών που δεν ε, εμπλέκονται με κάποιο τρόπο αλλά εξακολουθούν να αρνούνται το τι συνέβη από τον σύντροφό τους ακόμη και μετά την καταδίκη. Νομίζω λοιπόν ότι ίσως να πρέπει λίγο να εκπαιδεύσουμε και την κοινή γνώμη με κάποιο τρόπο. Όχι για να υποπτεύονται τους πάντες, αλλά εν πάση περιπτώσει για να γνωρίζουν ε, έτσι κάποια σημάδια ανησυχητικά ή προειδοποιητικά και να, γίνονται, να υπάρχουν κάποιες διαδικασίες ελέγχου κάθε τόσο ώστε να είναι και πιο εύκολο και για τα παιδιά να μιλήσουν. Και κάτι τελευταίο. Για αυτούς που ε, είναι θύματα ε, κακοποίησης μέσα από το κομπιούτερ, ας ελέξουμε και τα κομπιούτερ των παιδιών μας. Ε, εντάξει, λίγο συγκεχημένο όλα αυτά που είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτά, πρόεδρε, από μένα. Ευχαριστώ. αν κατάλαβα καλά την ερώτησή σας, αν γνωρίζουν οι δράστες ότι ε, βάζουν το υλικό στο ίντερνετ, ε, προφανώς το γνωρίζουν, ε, ε, αφού οι ίδιοι το βάζουν στο ίντερνετ. Εννοείται ότι και, φυσικά ξέρουν ότι υπάρχει και κόσμος που δεν θέλει να μπει σε αυτές τις ιστοσελίδες αλλά που με κάποιο τρόπο φτάνει σε αυτή την ιστοσελίδα ε, όχι, δεν ρωτούσα αυτό. Απλώς ρώτησα αυτοί που φτιάχνουν τις ιστοσελίδες, αυτοί που παρέχουν την ιστοσελίδα. Και νομίζω κάνατε ένα διαχωρισμό αυτών που βάζουν τις εικόνες στην ιστοσελίδα και αυτοί που, παράσχουν, που παρέχουν την ιστοσελίδα. Δεν ε, γνωρίζω εγώ απολύτως πώς, ποιος παρέχει το μηχανισμό για να δημιουργηθεί στο ιστοσελίδα ώστε να κυκλοφορήσετε το υλικό. Δηλαδή υπάρχει πιθανότητα αυτοί που διαχειρίζονται την ιστοσελίδα να είναι αθώοι ε, ε, σε σχέση με το υλικό που υπάρχει στην ιστοσελίδα που διαχειρίζονται. Δεν μιλώ για τους δράστες. Προφανώς οι δράστες δεν είναι αθώοι. Ίσως ε, εγώ δεν το, δεν το γνωρίζω. Ναι, να σας απαντήσω. Ε, κάποιες φορές ναι και κάποιες φορές όχι. Γιατί αν ας πούμε υπάρχει ένα web hotel προφανώς δεν ξέρεις ε, ακριβώς τι γίνεται και ποιος ανεβάζει υλικό ε, στο, στην ιστοσελίδα. Αλλά αν ξέρεις ότι υπάρχει αυτό το υλικό, τότε ναι, αν δεν κάνεις κάτι για να το κατεβάσεις, είσαι υπεύθυνος. Δηλαδή, ίσως κάποιος να είναι απλώς απρόσεκτος και να μην ελέγχει τι βάζει ο πελάτης του στην ιστοσελίδα. Ναι. Ε, εντάξει, δεν ξέρω αν μπορούμε να το πούμε απρόσεκτο, εν πάση περιπτώσει όμως, ε, ναι. εκουσίως είναι υπεύθυνο αν μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Οι providers στη Γερμανία που προσφέρουν δυνατότητες αποθήκευσης στο ίντερνετ δεν υποχρεούνται να ελέγχουν ενεργά αν μιλούμε για ποινικό υλικό ή όχι. Αν όμως το γνωρίσουν πρέπει να δράσουν. Αλλά αν δεν γνωρίζουν τι υλικό είναι αυτό και απλώς είναι παθητική πάροχη των υπηρεσιών, τότε δεν έχουν ευθύνη. Βέβαια αυτό είναι διαφορετικό σε κάθε χώρα. Όπως είπε και ο συνάδελφο, και ναι και όχι στην απάντησή σας. Υπάρχουν και κάποια μαύρα πρόβατα τα οποία ξέρουν ακριβώς τι, βάζουν στις, ε, τι αποθηκεύεται στις ιστοσελίδε τους. Υπάρχουν όμως και οι μεγάλοι πάροχοι ε, ίντερνετ που προφανώς δεν ξέρουν τι ακριβώς αποθηκεύεται στι ιστοσελίδε που προσφέρουν. Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να περάσουμε τώρα στο επόμενο πάνελ. Θα ήθελα λοιπόν να ζητήσω από τους ε, προσκεκλημένους μας να έρθουν εδώ στο Προεδρείο, την κυρία Τιάννα Σάτον, τον Πίτερ Ρόμπινς, τον Τζο Μακναμί, ο οποίος λείπει, τον Τζον Καρ,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 Λοιπόν, να ξεκινήσουμε το δεύτερο γύρο. Πρώτη ομιλήτρια η κυρία Διάννα Σάτον, η οποία εκπροσωπεί το NSPCC Αγγλίας. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Αντιπρόεδρε διότι δίνεται στην NSPCC την ε, δυνατότητα να πει κάποια πράγματα και να σας πούμε και εμείς γιατί θεωρούμε ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ σημαντικό βήμα για την προστασία των παιδιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Εθνική Εταιρεία για την Πρόληψη της Βίας στα Παιδιά είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός 126 χρόνων πείρας σε θέματα προστασίας παιδιών. Θέλουμε να μην υπάρχει βία στα παιδιά και συνεργαζόμαστε στενά με ε, ευρωπαϊκές μη κυβερνητικές οργανώσεις αντίστοιχου ε, ε, αντίστοιχου θέματος και ασχολούμαστε με θέματα σεξουαλικής κακοποίησης και σεξουαλικής εκμετάλλευσης πανευρωπαϊκά. Γιατί είναι σημαντική η νομοθεσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Από τα όσα γνωρίζουμε εμείς σε εθνικό επίπεδο, να γνωρίζουμε ότι πολλές πτυχές της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και κακοποίησης ε, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι έχουμε μεγαλύτερη μετακίνηση ε, ανά τον κόσμο και το κόσμο του ανάπτυξη του κόσμου του διαδικτύου ε, καταλαβαίνουμε ότι αλλάζει η ε, εθνική διάσταση και δεν μπορεί κάθε χώρα να δράσει μόνη της. Υπάρχει ευρωπαϊκή και παγκόσμια διάσταση. Γι' αυτό ακριβώς και χαιρετίζουμε την πρόταση για μια ευρωπαϊκή οδηγία. Ε, σύντομα θα ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε εδώ <laughs> ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη έχουν διάφορες υποχρεώσεις που προκύπτει από διεθνές δίκαιο για τα ανθρώπινα δικαιώματα ε, και πρέπει να διασφαλίσουν ότι τα παιδιά είναι η βασική μέρημνα σε όλες τις πτυχές της πολιτικής. Όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν κυρώσει την ε, ε, δήλωση για τα ε, τη Σύμβαση συγγνώμη, για τα Δικαιώματα των Παιδιών και το άρθρο 3 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επίσης και το άρθρο 24 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, δημιουργεί την υποχρέωση να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά προστατεύονται. Αυτό που κάνει οδηγία είναι το εξή. Προσπαθεί να αντιμετωπίσει κάποια από τα κενά που υπάρχουν στο παρόν νομοθετικό πλαίσιο και κυρίως ε, η απόφαση για την καταπολέμηση της σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών και τη παιδική πορνογραφία ήταν ένα πρώτο βήμα για να ενισχύσουμε την ε, συνεργασία και να προσπατατεύσουμε τα παιδιά από τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση. Ωστόσο, οι εκθέσει Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη μεταφορά τη οδηγία καταδεικνύουν ότι η απόφαση πλαίσιο περιλαμβάνει πολλά κενά και θα πρέπει φυσικά να προλάβει και τι εξελίξει, κυρίω ε, για το διαδικτυακό περιβάλλον. Όπω για παράδειγμα η αυξημένη χρήση του διαδικτύου από τα παιδιά, που φυσικά δημιουργεί και απελέ και ευκαιρίε. Επιπλέον, η οδηγία του 2003 εστιάζεται στην ε, τιμωρία των εγκλημάτων κατά παιδιών και επίσης θα πρέπει να περιλαμβάνουμε όμως και μέτρα για την πρόληψη των εγκλημάτων αυτών. Κυρίως ε, τα νέα άρθρα 27 και ε, συγγνώμη, 17 έως 19 της ε, πρότασης οδηγίας επειδή δεν έχω πολύ χρόνο και πολλά τα είπαν οι προλαλήσαντες, θα ήθελα να βασιστώ, ε, να μιλήσω κυρίως συγγνώμη για ένα ε, μέτρο πρόληψης ε, που αναφέρεται και στο άρθρο 10 της οδηγίας. Μας χαροποιεί το γεγονός ότι η οδηγία αναφέρεται στο γεγονός ότι θα πρέπει να καταγράφονται στο ποινικό μητρό κάποιου τα εγκλήματα κατά παιδιών και να υπάρχει ευρωπαϊκή ενημέρωση από αυτού, αλλά θεωρούμε ότι θα πρέπει να αναφέρονται και θέματα ε, ανθρώπων που απασχολούνται με παιδιά όταν έχουν τακτικές επαφές με παιδιά. Γιατί θεωρούμε ότι είναι σημαντικό αυτό. τα οποία ε, είναι παιδόφιλοι, ε, κάνουν πολλές φορές προσπάθειες για να βρίσκονται κοντά στα παιδιά. Όπως για παράδειγμα να ζητούν θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με παιδιά. Ε, η σεξουαλική βία διαπιστώθηκε μια έκθεση ε, ότι τις περισσότερες φορές είναι αποτέλεσμα ε, ανθρώπων που βρίσκονται στο οικογενειακό περιβάλλον των παιδιών ή άτομα εμπιστοσύνης. Ε, οι δάσκαλοι, οι εκπαιδευτές σε αθλήματα, αστυνομικοί και ούτω καθεξής. και υπάρχει ελάχιστη μέρημνα για το θέμα αυτό στην απόφαση πλαίσιο του 2003. Δεν υπάρχει καμία υποχρέωση για τους εργοδότες να ελέγχουν το ποινικό μητρό των ε, ατόμων που προσλαμβάνουν και δεν ανταλλάζονται αρχεία τέτοιων θεμάτων μεταξύ κρατών μελών. Θεωρούμε ότι τα θέματα της απασχόλησης είναι μια πολύ σημαντική δικλίδα ασφαλείας για να προστατεύσουμε τα παιδιά κατά της ε, κακοποίησης. Ε, εργοδότες ε, θα πρέπει να διαπιστώνουν αν υπάρχουν προηγούμενες κατεδίκες ώστε ε, τα άτομα αυτά να μην μπορούν να εργαστούν με παιδιά ή αν υπάρχει απαγόρευση σε εργασία με παιδιά. Επίσης, θα πρέπει να γίνονται οι ίδιοι έλεγχοι όταν κάποιος προσπαθεί να εργαστεί σε θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν με επαφή με παιδιά. Και αυτό θα πρέπει να γίνει και για ανθρώπους που έχουν ε, ζήσει στο εξωτερικό, διότι αυτή είναι η μεγαλύτερη πρόκληση αυτή τη στιγμή. Το να πρέπει να ελέγξει κάποιο αν έχει ποινικό μητρό κάποιο στι χώρε τι οποίε έζησε είναι αρκετά δύσκολο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό διότι ε, πολλοί εκμεταλλεύονται ακριβώ αυτό το δικαίωμα να μετακινούνται στα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταβαίνουν αλλού. Από τα στοιχεία που έχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο, 17.000. Ε, οι πίκοοι των νέων χωρών μελών ήρθαν στη Βρετανία από το 2004 και έκαναν αίτηση να εργαστούν σε, θέ, ε, σε θέσεις εργασίας που έχουν να κάνουν σε επαφή με παιδιά. Το 2004 μπορεί να γνωρίζετε την υπόθεση του Michael Forney που δείχνει τι ακριβώς μπορεί να συμβεί αν έρθει κάποιος από το εξωτερικό να εργαστεί που δεν, ε, στον οποίο δεν γίνεται κατάλληλος έλεγχος. Ο Φόρνι Ρέι πριν μετακομίσει στο Βέλγιο είχε αρκετές καταδίκες. Οι βελγικές αρχές φυσικά δεν γνώριζαν αυτές τις καταδίκες και ξεκίνησε να εργάζεται σε ένα σχολείο και φυσικά εκμεταλλεύτηκε τη θέση του για να κακοποιήσει σεξουαλικώς παιδιά. Το 2007 το NSPCC εξέδωσε μία έκθεση για την προστασία των παιδιών, την καλύτερη απασχόληση για τους εργαζομένους και διαπίστωσε στην έκθεση αυτή ότι τα άτομα τα οποία διαπράττουν σεξουαλικά δικήματα κατά παιδιών όλο ένα και πιο συχνά μεταφέρονται από τη μία χώρα στην άλλη καταδικασμένοι για σεξουαλικά δικήματα ε, ορισμένες φορές εκμεταλλεύονται τις διαφορές που υπάρχουν στα νομικά συστήματα των χωρών μελών και σε ορισμένες χώρες μέλη είναι πολύ πιο εύκολο να υπάρχει πρόσβαση σε θέσεις εργασίας με παιδιά από ό,τι σε άλλες χώρες. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει συνεργασία ώστε να διασφαλίσουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν θα εργάζονται με παιδιά όταν θα μετακομίσουν σε μια νέα χώρα. Και θα πρέπει να αναλάβουμε δράση τώρα, δεδομένου ότι γνωρίζουμε πράγματα και πρέπει να προσπαθήσουμε να ελαχιστοποιήσουμε του κινδύνου για τα παιδιά. Υπάρχουν μια σειρά από πρωτοβουλίε που θέλουν να αντιμετωπίσουν τη σεξουαλική κακοποίηση και τη σεξουαλική εκμετάλλευση και αυτά θα πρέπει να αποτελέσουν βάση για περαιτέρω συνεργασία, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι ε, δεν θα εργάζονται κατάλληλα άτομα με παιδιά ε, ακριβώς και μόνον επειδή μετακομίζουν σε μια άλλη χώρα. Θα πρέπει λοιπόν να γίνεται ανταλλαγή στοιχείων ποινικού μητρώου ε, και οι εργοδότες συχνά πρέπει να ε, προσπαθήσουν να αποκτήσουν πρόσβαση ποινικών μητρών από χώρε στι οποίε είναι πολύ δύσκολο, διότι κάποιε χώρε δεν δίνουν ποινικά μητρό, αντίγραφα ποινικού μητρό για αυτό το σκοπό. Όταν ληφθούν οι πληροφορίε, ορισμένε φορέ μπορούν να χρησιμοποιηθούν με δύσκολο τρόπο, γιατί ε, είναι γραμμένα σε άλλη γλώσσα ή αναφέρονται σε νομικού όρου που δεν μπορεί κάποιο να ερμηνεύσει και μπορεί ο εργοδότη να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει καταλήλω. Και επίση υπάρχουν ε, διαφορετικοί κανόνες αποθήκευση δεδομένων και εφαρμογή και αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην δίδονται κάποια στοιχεία. Επίσης, ορισμένες φορές ο νομικός ορισμός του ίδιου αδικήματος ε, είναι διαφορετικός και φυσικά αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν προβλήματα σε καταδίκες σεξουαλικών εγκλημάτων ε, κατά παιδιών. Ορισμένες φορές οι εργοδότε δεν μπορούν να αντιληφθούν τι ακριβώ λένε οι πληροφορίε και να κατανοήσουν αν υπάρχει κίνδυνο ε, για αυτού του ανθρώπου όταν εργάζονται με παιδιά. Είναι πολύ σημαντικό επίση τα κράτη-μέλη να έχουν ένα σύστημα για να χρησιμοποιούν τα ποινικό μητρώα ώστε να είναι βέβαιοι ότι ε, όσοι έχουν διαπράξει τέτοια εγκλήματα δεν θα εργάζονται με παιδιά και είναι πολύ σημαντικό λοιπόν ε, να υπάρχει καλή συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών. Συνοψίζοντα χαιρετίζουμε την υποχρέωση να γίνεται ανταλλαγή ή ποινικών μητρών όταν ετούνται ε, βάσει τη οδηγία, αλλά δυστυχώ δεν υπάρχει υποχρέωση να ελέγχεται κατά πόσον κάποιο εργάζεται ή έχει πρόσβαση σε παιδιά. Θα ήθελα τώρα εν συντομία να σταθώ και σε κάποια άλλα σημεία παρά το γεγονός ότι ε, οι άλλοι συνάδελφοι θα αναφερθούν στα θέματα αυτά. Καταρχάς, η συζήτηση για τον ορισμό του παιδιού. Αυτό ορίζεται σαφώς σε πολλά εφιστάμενα νομικά ε, κείμενα. Για παράδειγμα, στο άρθρο 2 για τα ανθρώπινα δικαιώματα της Σύμβασης ε, ε, του ΟΗΕ και υπάρχει και η ε, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Επίσης δεν θα πρέπει να γίνεται σύγχυση μεταξύ της ενηλικίασης και της ηλικίας συγκατάθεσης, η οποία είναι διαφορετική σε διάφορες χώρες. Επίσης Ε, μιλάμε πολύ συχνά για τις εικόνες ε, των παιδιών που είναι μία ε, απεικόνηση σεξουαλικής κακοποίησης που δημιουργεί πολύ περισσότερο πρόβλημα στα παιδιά διότι τα παιδιά γνωρίζουν ότι αυτή τη στιγμή έχει αναρτηθεί μία εικόνα στο διαδίκτυο μπορεί κάποιος να τη δει και να την κατεβάσει απεριόριστες φορές. Ε, θεωρούμε λοιπόν ότι το υλικό αυτό θα πρέπει να διαγράφεται, αλλά δυστυχώς η ταχύτητα με την οποία ε, κατεβαίνουν αυτές οι ιστοσελίδες ε, πρέπει να βελτιωθεί και θα πρέπει να μπλοκάρεται η πρόσβαση σε ιστοσελίδε που έχουν εικόνε σεξουαλικής κακοποίηση και βίντεο αντίστοιχα. Τέλος, το άρθρο 6, η ποινικοποίηση του grooming. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει σχετική οδηγία από το νομοθεσία συγγνώμη, από το 2003 και ε, βάσει αυτής της νομοθεσίας ε, έχουν εξοικειωθεί περισσότερα τα παιδιά γιατί γνωρίζουν τι ακριβώς σημαίνει και προσπαθούμε να ε, είμαστε και σε εγρήγορση και να προλαβαίνουμε τι τεχνολογικές εξελίξεις. Ελπίζουμε να μπορέσουμε να ε, προχωρήσουμε το κείμενο αυτό και να υιοθετηθεί αυτό το φιλόδοξο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος Ρόμπινς, ο οποίος εκπροσωπεί το Internet Watch Foundation. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Με καλέσατε για να αναφέρω την εμπειρία του Ηνωμένου Βασιλείου ως προς τα μέτρα μπλοκαρίσματος των σελίδων διότι η οργάνωσή μου αυτήν την ε, δουλειά κάνει στο Ηνωμένο Βασίλειο και καταρτίζει και κατάλογο ιστοσελίδων που εκμεταλλεύονται παιδιά σεξουαλικώς. Η κατάρτιση αυτών των μητρών και το μπλοκάρισμα είναι τα κύρια μέτρα που παίρνουμε ώστε να συμπληρώνουμε τη δουλειά των δικαστικών αρχών και άλλων που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν την κακοποίηση των παιδών. Βέβαια πάντα συμβαίνει κάποια καθυστέρηση από τη στιγμή που παίρνετε μια απόφαση μέχρι να εφαρμοστεί. Υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ότι είναι αποτελεσματική η κατάρτιση του Μητρώου και το μπλοκάρισμα. Πριν από δύο χρόνια όταν πρωτοκαταρτίζαμε τον κατάλογό μας υπήρχαν πάνω από 1500, 1500 κλήσεις τέτοιων σελίδων την ημέρα και σήμερα έχει μειωθεί σε 800 ευρωώρες την ημέρα. Σήμερα δε το πρωί μάθαμε ότι 400 ιστοσελίδες έχουν καταγραφεί ως παιδική πορνογραφία και λίγες μόνο από αυτές είναι παλαιότερες από ένα μήνα. Άρα τα μέτρα μπλοκαρίσματος έχουν αρχίσει να αποδίδουν αυτό. Καταλαβαίνω εγώ. Το Internet Watch Foundation βέβαια δεν είναι δημόσια υπηρεσία ε, εργάζεται σε συνεργασία με τους προμηθευτές κατασκευαστές κινητών, φορητών τηλεφώνων κλπ. κλπ. Είναι ιδιωτική. Και συνεργαζόμαστε και διεθνώς με το HOPE και άλλα, άλλες διεθνείς οργανώσεις για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα από το 1996. Πάνω από 300.000 αναφορές έχουμε διεκπαιρεώσει για να δούμε ποιες είναι οι τάσεις που παρατηρούνται στον κυβερνοχώρο. Η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών από το ίντερνετ έχουμε θελήσει να δούμε αν αποδίδει χρηματικά. Δεν υπάρχουν στοιχεία σίγουρα αλλά προσπαθούμε να δούμε ποια είναι η τεχνική που χρησιμοποιούν οι παραβάτες τεχνική η οποία όλο και πιο πολύπλοκη γίνεται. Οι προμηθευτές και όσοι διανέμουν τέτοιο υλικό προσπαθούν με κάθε τρόπο να διαδώσουν το υλικό αυτό παρακάμπτοντας έτσι την λίγη νομοθεσία που ισχύει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν δίκτυα ιστοσελίδων που ανακαλύπτουν όλο και πιο καινούργιες μεθόδους για πληρωμές και για διεθνή συνεννόησή τους. Και προσπαθούν επίσης να επιταχύνουν τις υπηρεσίες αυτές για να αποφύγουν έτσι την ταύτισή τους από τις υπηρεσίες δίωξης. Είναι δύσκολο να φανταστούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουν στο μέλλον τα μέτρα που υπάρχουν, αλλά είναι σίγουρο ότι κάτι θα βρουν. Προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε έρευνες πιο μακροχρόνιες και σε διεθνή συνεργασία για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Είναι ουσιώδες, όποιος παίζει κάποιο ρόλο και θέλει να είναι πιο ασφαλές στο ίντερνετ να γνωρίζει ότι πρέπει να αντιμετωπίσει και το πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν πολλά κόλπα που χρησιμοποιούν οι παραβάτες αλλά και πολλοί τρόποι αντιμετώπισης. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει διεθνής συμφωνία και συνένεση για την τακτική που πρέπει να ακολουθηθεί. Μερικές χώρες, από ό,τι ξέρουμε, δεν έχουν κανένα καθορισμένο σύστημα για, την, για το κλείσιμο τέτοιων ιστοσελίδων. Και συνεχίζεται η συζήτηση σε μερικές χώρες, δεν ξέρουν ακόμη ποιος έχει την ευθύνη, ποιος μπορεί Ποιος έχει τη δυνατότητα να κλείσει μια ιστοσελίδα. Ιδεοδός θα έπρεπε να υπάρχει μία διεθνής υπηρεσία διοκτική που να ασχολείται μόνο με αυτό. Γιατί δεν μπορούν να λυθούν όλα αυτά τοπικά ή εθνικά. Γενικά υπάρχει συμφωνία ότι πρέπει να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά από την κακοποίηση και να διωχθούν οι χρήστες. Δεν υπάρχει συμφωνία ως προς το πώς ακριβώς μπορεί και πρέπει να γίνει αυτό. Εξάλλου το περιεχόμενο των ιστοσελίδων παραμένει διαθέσιμο ακόμη και αν υπάρχει κάποια διοκτική διαδικασία. Το μπλοκάρισμα ιστοσελίδων είναι μια ιδέα που έχει συζητηθεί εδώ και πολλά χρόνια και εμείς καταρτίζουμε ένα κατάλογο που να διευκολύνει την ε, πρακτική αυτή. Ο κατάλογος αυτός βέβαια καταρτίζεται εθελοντικά με βάση 60 εταιρείε στο Ηνωμένο Βασίλειο και διεθνώς. 98,6% των ε, ταχαίων διασυνδέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο χρησιμοποιούν τον κατάλογό μας. Στο Ηνωμένο Βασίλειο ζητούμε όταν ταυτιστεί κάποια τέτοια ιστοσελίδα την άμεση, το άμεσο μπλοκάρισμά της. αλλά αυτό δεν μπορεί να γίνει παρά μόνο και με διεθνή συνεννόηση ώστε να μην μεταφερθεί αμέσως αλλού η ιστοσελίδα αυτή. Οι εικόνες που εξετάζουμε σύμφωνα με την ομοθεσία του Ηνωμένου Βασιλείου ταξινομούνται σύμφωνα με τα κριτήρια που έχουν καθορίσει δικαστέ. Η διευκόλυνση του μπλοκαρίσματος είναι κάτι πολύ χρήσιμο και τη δουλειά μας την ελέγχει και ανεξάρτητος οργανισμός. Ακολουθούμε νομικές συμβουλές από ειδικού επιχειρήσεων, από οικευμένους αστυνομικούς, ώστε να είμαστε βέβαιοι ότι αυτά που κάνουμε συμφωνούν απόλυτα με την ισχύουσα νομοθεσία. Η ταξινόμηση λοιπόν και η κρίση του περιεχομένου μιας ιστοσελίδα και η ένταξη στον κατάλογο γίνονται με αυστηρά κριτήρια. Τονίζω ότι δεν έχουμε καμία δικαιοδοσία για δίωξη των παραβατών μόνο το περιεχόμενο εξετάζουμε. Οι περισσότερες αναφορές που εξετάζουμε αφορούν βέβαια υλικό που έχει αναρτηθεί στο εξωτερικό και δεν έχουμε πολλές δυνατότητες να αντιδράσουμε. Ούτε χρηματοδοτούμαστε από την κυβέρνηση της χώρας, του Ηνωμένου Βασιλείου, και προφανώς δεν έχουμε κανένα κέρδος. Οι περισσότερες ιστοσελίδες της αστυνομίας λένε στο κοινό να απευθυνθεί σε Θεωρούμε όμως ότι οι κατάλογοι πρέπει να αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Γιατί αλλιώς δεν πρόκειται να έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Από ό,τι γνωρίζουμε η σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών είναι κάτι που αλλάζει συνεχώς και για να είμαστε συνοπτικοί και να αποφύγουμε την, το άχρηστο μπλοκάρισμα απαρχαιωμένων και άχρηστων ιστοσελίδων πρέπει συνεχώς τουλάχιστον μία φορά τη μέρα να τα ενημερώνουμε όλα αυτά τους καταλόγους. Το μπλοκάρισμα κατ' εμάς πρέπει να γίνεται με τρόπο διαφανή και να εξυπηρετεί το ευρύτερο κοινό. Να υπάρχει ένας εύκολος τρόπος να ελέγξει ο πολίτης αν υπάρχει ή όχι μπλοκάρισμα και να εμφαίνεται αυτό μόλις κάποιος ζητήσει μια ιστοσελίδα. Επίσης πρέπει να υπάρχει η δυνατότητα οποιοδήποτε έχει αντίρρηση για κάποιο περιεχόμενο να παραπονεθεί και να ζητήσει περίληψη της στο σελίδα στο κατάλογο. Έχουν ακουστεί ανησυχίες ότι οι υποδομές που διευκολύνουν το μπλοκάρισμα μπορεί να τύχουν κατάχρησης από εγκληματίες. Πρέπει λοιπόν να υπάρξουν εγγυήσει ώστε να ελαχιστοποιηθεί αυτή η πρακτική και να διατηρηθεί ταυτόχρονα το μπλοκάρισμα. Στο Ηνωμένο Βασίλειο τα έξι χρόνια που ασχολούμαστε δεν έχει υπάρξει κανένα τέτοιο πρόβλημα. Επειδή είναι σχετικά μικρό το ποσοστό των ιστοσελίδων παιδικής πορνογραφίας, πρέπει το τα μέτρα που λαμβάνουμε για το μπλοκάρισμα να, είναι, να μην είναι δυσανάλογα με την παράβαση. Κανείς όμως δεν πρέπει να έχει το δικαίωμα πρόσβαση σε παιδική πορνογραφία και άρα το μπλοκάρισμα αν γίνεται με έξυπνο τρόπο μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό μέτρο καταπολέμησης. Και τέλος, η χορήγηση του καταλόγου σε μια εταιρεία δεν εγγυάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και η εταιρεία και την ενημέρωση που πρέπει να έχει τακτικά. Γι' αυτό η μέθοδη πιστοποίησης της αποτελεσματικότητας της χρήσης του καταλόγου είναι κάτι που το ψάχνουμε ακόμη. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο λόγος στον Τζον Μακναμή, ο οποίος εκπροσωπεί τη European Digital Rights. Παρακαλώ. Ευχαριστώ που μου δίνετε και τον λόγο και την ευκαιρία να μιλήσω και εγώ για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα. Η European Digital Rights είναι μια ένωση 27 ε, ε, ενώσεων ε, πολιτικών δικαιωμάτων από τα κράτη μέλη της Ένωσης. Δουλεύω εδώ και ένα χρόνο στην εταιρεία αυτή και πριν ασχολήθηκα εντατικά με τον τομέα του ίντερνετ και της τεχνολογίας. Ένα σημείο θα ήθελα εγώ να θίξω μέσα σε αυτή την τεράστια οδηγία, το, η φραγή το, των ιστοσελίδων στο ίντερνετ. Και θα ήθελα επίσης να πω για να μην παρεξηγηθώ ότι αυτό είναι ένα τμήμα μιας μεγάλης οδηγίας. Η, τα κριτικά μου σχόλια για το ένα άρθρο αυτό δεν, σημαίνουν, σημαίνουν ότι είμαι επικριτικός αντί όλες τις οδηγίες. Τέσσερα σημεία θα ήθελα να αναφέρω. Ε, δεκαπέντε θα ήθελα να σας αναφέρω, αλλά μόνο δέκα λεπτά έχω. Οπότε θα ξεκινήσω. Η φραγή δεν βοηθά στο να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα, γιατί αποτελεί μεγάλο κίνδυνο και για την κοινωνία και για το ίδιο το παιδί και για την προστασία του. Η Κομισιόν κάνει την πρότασή της, αλλά χωρίς να έχει κάνει σωστή ανάλυση και η πρόταση της Κομισιόν ε, για να περιοριστεί το μπλοκάρισμα μόνο σε, σε σελίδες ε, ε, παιδικής, παιδικής προγραφίας δεν έχει τηρηθεί. Καταρχήν, γιατί είναι επικίνδυνο αυτό. Η φραγή είναι γενικός όρος. Υπάρχουν διάφορα είδη φραγής. αυτή που, αυτό, η φραγή που κάνει το Internet Web Foundation είναι διαφορετική από τη φραγή που κάνουν οι Σουηδικές Αρχές, ας πούμε. Υπάρχουν δύο είδη φραγής. Ε, το πιο ε, σύνηθες είναι η, το να μπλοκάρονται σελίδες που ε, οδηγούν, είναι σαν σύνδεσμοι και οδηγούν σε σελίδες πορνογραφικού περιεχομένου. Και οδηγούν τους καταναλωτές στις σελίδες αυτές χωρίς ο καταναλωτής να έχει δώσει πρώτα τη σύμφωνη γνώμη του. Μιλούμε για μεγάλη δηλαδή έκταση και χρήση της ε, τεχνολογίας ε, μέσω της ε, εκμετάλλευσης ας των προσωπικών email των καταναλωτών αλλά και, πάλι το, μέσω της, του κωδικοποιημένου μηνύματος το πεδίο εφαρμογής αυτών των τεχνολογιών είναι πολύ περιορισμένο. υπάρχουν και πολύ λίγες αποδείξεις για το ποιο είδος φραγής περιμένει η Κομισιόν να εφαρμοστεί. Και μόλι εφαρμοστεί η οδηγία, η Κομισιόν δεν θα έχει και καθόλου έλεγχο στο ποια τεχνολογία θα χρησιμοποιήσουν τα κράτη-μέλη ω ε, την ε, καταλληλότερη. Οπότε η φραγή δεν δουλεύει. Γιατί όταν φράσονται οι, ε, οι ιστοσελίδε, αυτέ εξακολουθούν να είναι online. Πολλοί χρησιμοποιούν πάρα πολύ πάρα ενισχυμένη τεχνολογία που την υποστηρίζει η Κομισιόν για να ξεπεράσουν αυτή την φραγή η φραγή δεν αντιμετωπίζει τα προβλήματα της παιδικής κακοποίησης ε, που προκύπτουν μέσα από άλλες πλατφόρμες όπως η peer-to-peer και όπως είπε και ο κύριος από την, από την Σουηδία ε, υπάρχουν και άλλες ε, και άλλοι λόγοι τους οποίους η φραγή είναι αναποτελεσματική. Οπότε το πεδίο που έχουμε για να χειριστούμε το θέμα μέσω της φραγής είναι πολύ περιορισμένο. Ούτε η τυχαία ε, πρόσβαση είναι, περιορίζεται μέσα τη φραγή. Μόνο ένας ανά τρεις χιλιάδες αναφέρουν ότι έχουν ε, ε, βρεθεί κατά λάθο σε μια τέτοια παράνομη ιστοσελίδα. Βεβαίω αυτό μπορεί να βοηθήσει και τι εμπορικέ σελίδε, γιατί μόλι δουν ότι έχουν μπλοκαριστεί, μπορούν να πάνε σε άλλο σερβερ, σε άλλη χώρα και να συνεχίσουν τι δραστηριότητέ του η ε, ε, με τη φραγή παραμένουν λοιπόν online στους σελίδες και δεν βοηθά αυτό σε τίποτα. Δεύτερον, ο κίνδυνος για το παιδί, για την προστασία του και για την κοινωνία. Υπάρχουν διάφορα είδη κινδύνων που προκύπτουν από τη φραγή, από την, για την προστασία των παιδιών, για την ε, διεθνή εξοπιστία της Ένωσης και για την ασφαλεία της κοινωνίας. Ήδη έχουμε πολλούς ανθρώπους που, που δημιουργούν ε, τις χειρότερες δυνατές ε, λίστες αντί να αντιμετωπίζουν πραγματικά το πρόβλημα. Υπάρχουν πάρα πολλές ε, ιστοσελίδες που συνήθως βρίσκονται στις, παρέχονται μάλλον από τους μεγάλους εμπορικούς παρόχους ίντερνετ. Προσπαθούμε λοιπόν και σε διεθνέ επίπεδο να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Ε, Επίση, το μπλοκάρισμα ε, παραλύει λίγο τα κρατημέλη και δεν τα αφήνει να δράσουν άμεσα. Η Κομισιόν ε, είπε ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει αυτή η οδηγία, λέγοντα ότι δεν μπορούμε να επικιστευτούμε τα κρατημέλη για να εφαρμόσουν την σύμβαση του Συμβουλίου τη Ευρώπη άμεσα ή σωστά. Και σε τέτοιε συνθήκε το χειρότερο που μπορεί κανεί να κάνει είναι να προωθήσει ένα μέτρο που επιτρέπει στα κρατη να ε, κρύψουν την ε, ανεπάρκειά του. Και αυτό ακριβώ έγινε. Αν ε, το μπλοκάρισμα δείχνει ότι κάτι γίνεται για την αντιμετώπιση τη παιδική προγραφία online, ξέρουμε ότι θα μειωθεί η πίεση για να άλλα πιο αποτελεσματικά μέτρα. Και οι πόροι θα δοθούν σε άλλους, σε άλλους τομείς που επίσης πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα. Και το πρόβλημα επίσης ε, έχει να κάνει και με το μπλοκάρισμα άλλων τομέων, ε, που το βλέπουμε και σε, κράτη, σε άλλα κρατημέλη. Ήδη το μπλοκάρισμα χρησιμοποιείται για, να, ε, για, να για, να, για το τζογάρισμα online και για άλλες δραστηριότητε. Υπάρχει επίσης και κόστος προς την τεχνολογία, γιατί θα χρειάζονται πολύ περισσότερα τεχνολογίες για να υπάρχει πρόσβαση στο ίντερνετ το μπλοκάρισμα θα πλήξει την αξιοπιστία της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω του κολλήματος που θα υπάρχει στην ελευθερία ε, ενημέρωσης. Πώς μπορούμε λοιπόν να την ενισχύσουμε σε λίγα χρόνια, όταν θα έχουμε εφαρμόσει το, μια σωστή ε, αποτελεσματική δυνατότητα φραγής... ...όπως αυτή που κάνουμε για να μπλοκάρουμε τι τις ιστοσελίδε τζόγου, δείχνει ότι πραγματικά κρύβουμε την ανεπάρκειά μας. Υπάρχουν πολύ λίγε αποδείξει ανάλυση τη της που θα έχει όλο αυτό από την Κομισιόν στα κράτη-μέλη. Οι κίνδυνοι είναι πολλοί. Δεν μπορούμε να εφαρμόζουμε και να χρησιμοποιούμε τεχνολογίε που, που δεν έχουν αποδειχθεί ότι είναι αποτελεσματικέ σε διεθνέ επίπεδο. Η, πρέπει να έχουμε πραγματικές, πραγματικά μέτρα και όχι απλώ συμβολικά. Η πρόταση αυτή περιλαμβάνει πολύ μεγάλου κινδύνου και για την προστασία των παιδιών και για την κοινωνία. Τρίτον, η δουλειά που γίνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Επιτροπή ξεκίνησε τις αξιολογήσεις επιπτώσεων για να αξιολογήσει τις, ε, ε, την συνεκτικότητα των οδηγιών της και να οδηγήσει σε ένα ε, σωστό ρυθμιστικό περιβάλλον. Η, ο τομέας αυτός όμως χρειάζεται και ποιότητα και συνεκτικότητα και αποτελεσματικότητα και απόδοση. Αλλά πώς, ε, αποτελε, πόσο, αποτελεσματικός, πόσο αποτελεσματική θέλει να είναι όντω η Κομισιόν προτείνοντας το υφραγή χωρίς να προσπαθήσει να ε, αξιολογήσει την επίπτωση σε χώρε όπου η υφραγή ήδη υπάρχει χωρίς να βλέπει κατά πόσο μπορεί να ε, υπάρξει διάλογος με άλλες χώρες, ε, όπως με τη ΣΥΠΑ για, τον, για το θέμα αυτό, χωρίς να αξιολογήσει συγκεκριμένα γιατί οι ιστοσελίδες αυτές παραμένουν online, ακόμη και όταν μπλοκάρονται. Και εδώ θα ήθελα να αναφέρω και την, το δελτίο τύπου από την Γερμανία, από το γερμανικό τύπο που έχει γίνει, αναφέρει μια ανάλυση που έχει γίνει από αυτού. Επίσης η Κομισιόν δεν έχει αναφέρει την, ε, σχετικότητα που υπάρχει και τις ε, αυξανόμενες ποσότητες πορνογραφικού υλικού που ε, υπάρχουν σε σερβερς ή σε διάφορες άλλες ιστοσελίδες. Και το ξενόμενο πρόβλημα επίσης ότι οι ιστοσελίδες ε, γρήγορα κινούνται, δηλαδή πολύ γρήγορα ε, δραστηριοποιούνται ώστε δεν μπορούν να μπουν στις, ε, στους διάφορους καταλόγους. Οπότε πού ακριβώς βάζουμε τη γραμμή της αναλογικότητας. Η Κομισιόν δεν είναι σαφή ό,τι αφορά το στόχο του εισφραγή, αν δηλαδή μιλούμε για ε, ε, πρόσβαση σε τέτοιε ιστοσελίδε ή αν πρόκειται για πρόσβαση ευκαιριακή. Υπάρχει μια ε, έκθεση από τον ΑΣΑ που λέει ότι είναι πολύ ε, μεγάλη η κίνδυνη ε, και δυνάμει της Ευρωπαϊκής Σύμβασης του, της για τα δικαιώματα του παιδιού μπορεί να, η προσέγγιση του Κομισιόν να, να αποδειχθεί παράνομη. Η Κομισιόν επίσης δεν έθιξε το θέμα αυτό ούτε σε επίπεδο επικουρικότητας. Όλα αυτά λοιπόν έχουν τεράστιες συνέπειες και ο κίνδυνος όλων αυτών των συνεπειών είναι υπαρκτός. Για παράδειγμα, όπως πολλοί που μίλησαν σήμερα, ε, το λόμπι της Δανίας για την πνευματική διοκτησία ε, απαιτεί να μπλοκαριστούν κάποιες ιστοσελίδες και είπαν ότι έπρεπε να δει ο κόσμος ότι κάνουμε κάτι. Χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα ή τις συνέπειες ή την αναλογικότητα, δόθηκε η εντολή και η κυκλοφορία σε αυτή την ιστοσελίδα αυξήθηκε αμέσως κατά 12%. Η ε, διαρροή λοιπόν τέτοιων ε, ιστοσελίδων συνήθως αυξάνει την κυκλοφορία και την επισκεψιμότητά τους. Επίσης, ε, το να πειραματιζόμαστε με μη, μη αποδεικτές ιστοσελίδες και τεχνολογίες είναι αναποτελεσματικό. Είναι ίσως και επικίνδυνο. και μόλις εφαρμοστεί θα είναι πολύ δύσκολο να, να καταργηθεί. Η Κομισιόν δεν έχει αξιολογήσει αν όντω το blocking θα μπορούσε να ενισχύσει τις ιστοσελίδες αυτές. Είδαμε πώ γίνεται η φραγή των ιστοσελίδων σε κάποιε κάποιες χώρε και δεν, η Κομισιόν δεν αξιολόγησε καν αν υπήρξε κάποια αξία μετά από αυτό. Αν δηλαδή όντω διεκόπηκαν τα μονοπόλια τζόγου μετά από τον μπλοκάρισμα των σχετικών ιστοσελίδων. Η Κομισιόν μα υποσχέθηκε ότι αυτό που γίνεται πια δεν θα γίνεται. Αλλά αυτό δεν μας λέει τίποτα. Η Κομισιόν υποστήριξε ότι θα, το μπλοκάρισμα θα γίνεται μόνο για ιστοσελίδε παιδική πορνογραφία. Ούτε αυτό ισχύει. Καλό θα ήταν να μπορούμε να πιστέψουμε τι ε, υποσχέσει τη Κομισιόν. Παρ' όλα αυτά, η ίδια η Κομισιόν ε, χρηματοδοτεί δύο προγράμματα που έχουν στόχο να μπλοκάρουν άλλο, ε, ιστοσελίδε με άλλο περιεχόμενο. Το Συμβούλιο η τελευταία προεδρία μάλλον, ε, υποστήριξε το συγκεκριμένο έγγραφο για την προστασία των ε, μονοπωλίων τζόγου σε χώρες όπως η Λιθουανία, η Ιταλία, η Γερμανία, η Γαλλία. Ε, έχουν τέτοιες συμφωνίες για να προστατευτούν τα μεγάλα εμπορικά συμφέροντα. Η υπόσχεση λοιπόν που μα δόθηκε από την Κομισιόν δεν τηρείται. Ναι. Ούτε από τα κρατημέλη, ούτε από την Κομισιόν, ούτε από το Συμβούλιο. Κλείνοντα, θα ήθελα να ενθαρρύνω την Επιτροπή σας να μελετήσει όλα τα θέματα αυτά και να ε, υποβάλει μια πρόταση που θα σέβεται το κράτος δικαίου και που δεν θα ε, ε, μετακυλεί την ευθύνη στα κράτη-μέλη, τα οποία τη μετακυλούν μετά σε τρίτους η οδηγία λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να δράσουν έναντι πραγματικών ε, εγκλημάτων. Δεν μπορούν να κρύβονται πίσω από την ανεπάρκειά τους και το, η, διάταξη που αφορά τη φραγή θα πρέπει να διαγραφεί, να αφαιρεθεί από την οδηγία. Πρέπει τα κράτη-μέλη επιτέλου να, κάνουν, να αναλάβουν αυτό που τους υποχρώνουν να κάνουν η σύμβαση που έχουν υπογράψει για τα δικαιώματα του παιδιού και η δήλωση από τη Στοκχόλμη και η ε, γενική ε, δήλωση που υπάρχει της Οκλαχώμα. Δεν μπορούμε να ακούμε πια κενές υποσχέσεις. Ευχαριστώ. Ε, Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα το λόγο έχει η Κριστιάνα Ντεπάολη η οποία εκπροσωπεί το Save the Children. Παρακαλώ. Χωρίς μικρόφωνο η ομιλήτρια. Sorry. Θα ήθελα να ευχαριστήσω εξ ονόματος ε, του Save the Children Ευρώπης που εκπροσωπώ σήμερα την κυρία Αντζελίλη και την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών και Εσωτερικών Υποθέσεων, διότι μα έδωσε τη διευκαιρία να μιλήσουμε σήμερα για την οδηγία για τη σεξουαλική κακοποίηση και εκμετάλλευση των παιδιών. Το Save the Children είναι η μεγαλύτερη ανεξάρτητη μη κυβερνητική οργάνωση για την προστασία των παιδιών ε, ιδρύθηκε το 1919, βρίσκεται σε πάνω από 118 χώρες στον, χρόνο και, ε, το, στον κόσμο και έχουμε ένα δίκτυο 18 ε, κεντρικών γραφείων και ένα κεντρικό γραφείο συντονισμού. Χαιρετίζουμε την πρόταση αυτή διότι προσπαθεί να βελτιώσει και να κάνει πιο αποτελεσματικό το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και σεξουαλική εκμετάλλευση των παιδιών. Παρ' όλα αυτά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να διασφαλίσει ότι θα ληφθούν αποτελεσματικά μέτρα και ε, όσο το δυνατόν υψηλότερα πρότυπα στι χώρε Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε οι ανήλικοι οι οποίοι είναι θύματα κατοικοποίηση, καταρχά να εντοπίζονται και από εκεί και πέρα να ε, την χάνουν τη ε, υποστήριξη. Όλα αυτά φυσικά θα πρέπει να γίνονται βάσει των αρχών που ε, κηρύσσει ο ΙΕ στην ε, αρχή για τα δικαιώματα των παιδιών και στην αρχή που αναφέρεται στα συμφέρον των παιδιών. Το Save the Children προσπαθεί να δει την ε, οδηγία αυτή συνολικά και συνεργασία με άλλες κυβερνητικές οργανώσεις ε, οι οποίες είναι παρούσες εδώ ε, προσπαθήσαμε να κάνουμε κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις ε, διεξοδικές οι οποίες θέλουν να ε, προτείνουν κάποιες βελτιώσεις και κάποιες αλλαγές στο κείμενο και σε κάποια άρθρα της οδηγίας. Για λόγους χρόνου θα εστιάσω μόνο στα άρθρα τα οποία αναφέρονται κυρίως στην προστασία, στη συνδρομή και στην υποστήριξη των ανηλίκων θυμάτων από την πείρα μας γνωρίζουμε και νομίζω ότι το ακούσαμε και σήμερα το πρωί ότι η μεγαλύτερη πλειοψηφία των παιδιών ε, τα οποία είναι θύματα σιωπούν ακόμα και όταν ενηλικιώνονται για τα όσα του συνέβησαν. Οι λόγοι είναι διάφοροι, δεν υπάρχει ο χρόνο εδώ να επισέλθω σε λεπτομέρειε, αλλά απλώ να πω ότι τα ανήλικα θύματα πολλέ φορέ ε, υποχρεούνται στη σιωπή από τον ίδιο τον ε, άνθρωπο που του κακοποίησε, που πολύ συχνά είναι ένα πολύ κοντινό του άτομο, το οποίο εμπιστεύονται. Και πολλέ φορέ η κακοποίηση συνοδεύεται από αισθήματα ντροπή που φυσικά ε, ελαχιστοποιούν το ενδεχόμενο να ε, ομολογείς κάποιος τι του συνέβη. Προσπαθούμε λοιπόν να βρούμε τρόπους ε, να εντοπίζονται τα θύματα και μας χαροποιεί το γεγονός ότι υπάρχουν μέτρα στην οδηγία που οδεύουν προς αυτή την κατεύθυνση. Αναφέρομαι στο άρθρο 15 και θεωρούμε πολύ θετικό το γεγονός ότι λαμβάνονται μέτρα ώστε να ενθαρρύνονται τουλάχιστον όσοι έρχονται σε στενή επαφή με ανήλικα παιδιά να ε, καταγγέλουν οι υποθέσεις κακοποίησης. Και φυσικά ε, να τονίσουμε ότι θα πρέπει να υπάρχει και κατάλογη, κατάλληλη επιμόρφωση των ανθρώπων αυτών που θα τους επιτρέπουν να ερμηνεύσουν καταλήλως ε, τις ενδείξεις ε, μιας πιθανής κακοποίησης. Θεωρούμε πολύ θετικά τα μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται στο άρθρο 14 που θέλουν να κάνουν πιο αποτελεσματική την ερευνητική δουλειά των αστυνομικών δυνάμεων αλλά οι έρευνες που σχετίζονται με τις υποθέσεις σεξουαλικής κακοποίησης των παιδιών θα πρέπει να θεωρούνται προτεραιότητα, να μην υπάρχουν επικίνδυνες καθυστερήσει και να λαμβάνουμε πάντα υπόψη το συμφέρον των παιδιών. Ελπίζουμε και αυτή είναι και η περίπτωση των ε, σεξουαλικών κακοποίησεων των παιδιών για την ε, προστασία ε, υλικού παιδικού περνογραφίας ε, ότι θα υπάρξουν μέτρα τα οποία θα ενισχύσουν τη συνεργασία μεταξύ των χωρών και το συντονισμό μεταξύ των χωρών και σε διεθνές επίπεδο όσον αφορά τις ερευνητικέ του εργασίε και ελπίζουμε να υπάρξουν μέσα και αποτελεσματικές έρευνες όπως για παράδειγμα έρευνε οι οποίε θα γίνονται υποκάλυψη. υπογράμμισαν πολλοί από μεν, ε, πριν από μένα ότι θα πρέπει να ε, εντοπίζεται και το υλικό παιδικής πορνογραφίας, διότι πολλές φορές αυτό είναι και το υλικό που επιτρέπει να ε, γίνει δίωξη των εγκληματιών. Μας ε, αρέσει ιδιαίτερο το άρθρο 14.3 που ζητά από τα κράτη-μέλη να έχουν ερευνητικές, ε, ερευνητικά τμήματα τα οποία θα μπορούν να βοηθήσουν να εντοπίζονται οι ανήλικοι βάσει του υλικού αυτού και ε, θέλουμε να σας παρακινήσουν να υπάρχουν ανθρώπινοι αλλά και οικονομικοί πόροι προκειμένου να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε αποτελεσματικό διότι όπως ακούσαμε σήμερα το πρωί αυτά είναι πάρα πολύ περίπλοκα και πολύ δύσκολα πράγματα. Επίσης, το γεγονός ότι εισάγεται ως ε, ποινικά κολάσιμο αδίκημα το grooming ε, ε, θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό διότι προσπαθούμε να βρούμε τους διάφορους τρόπους με τους οποίους μπορεί κάποιος να παραπλανήσει έναν ανήλικο. Το άρθρο 6 αναφέρεται όμως στους ανήλικους κάτω από την ηλικία συγκατάθεσης. Για μας αυτό είναι ανησυχητικό διότι ε, είναι εκτεθειμένα και δεν προστατεύονται ε, τα ανήλικα παιδιά τα οποία έχουν φτάσει στην ηλικία συγκατάθεσης μεν αλλά δεν έχουν φτάσει στα 18. Γι' αυτό λοιπόν ε, θεωρούμε ότι θα πρέπει να διαγραφεί εδώ η ηλικία συγκατάθεσης. Ε, τέλος, το Save the Children θεωρεί θετικό το γεγονός ότι επικεντρώνεται στην προστασία των παιδιών και στη συνδρομή των θυμάτων η οδηγία αλλά θεωρούν ότι τα παιδιά θύματα θα πρέπει να ε, είναι αντικείμενο προσοχής και να λαμβάνονται υπόψη ε, το συμφέρον τους πάντα και τα δικαιώματά τους. Θεωρούμε θετικά τα μέτρα, αλλά ελπίζουμε ότι χάρη στη συζήτηση η οποία είναι εξελίξη, τα άρθρα 18 και 19 θα ενισχυθούν ώστε να περιλαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι τα κράτη-μέλη θα υιοθετήσουν εθνικές συστημικές στρατηγικές για την προστασία και υποστήριξη των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης και να υπάρχουν πειθαρχικές διαδικασίες κατά της κακοποίησης ώστε να μπορέσουμε να έχουμε συνεργασία και συντονισμό των ενδιαφερομένων φορέων, κυρίως των αστυνομικών δυνάμεων και των κοινωνικών υπηρεσιών, αλλά φυσικά και του δικαστικού συστήματος. Εν τέλει, θεωρούμε ότι είναι θετικό το γεγονός ότι δίνεται προσοχή ε, στα μέτρα προστασίας ε, των θυμάτων κατά τη διάρκεια της ε, δίκη και της ερευνητική και ανακριτικής διαδικασίας. Τα τραύματα τα οποία αντιμετωπίζουν τα παιδιά δεν θα πρέπει να επιδεινώνονται σε αυτό το στάδιο της διαδικασίας και θα πρέπει να διασφαλίσουν ότι το συμφέρον των ανηλίκων γίνεται πάντα σεβαστό. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει όλοι όσοι έρχονται σε επαφή με παιδιά να είναι κατάλληλα καταρτισμένοι και να γνωρίζουν τα δικαιώματα των παιδιών. Πέραν των μέτρων αυτών, ε, στην ε, σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την ε, εκμετάλλευση και την κακοποίηση περιλαμβάνονται και άλλα μέτρα τα οποία θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει και να λάβει υπόψη της κυρίως τον ορισμό ώστε να είναι τέλεια η εν λόγω οδηγία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα να καλέσουμε εδώ στο Προεδρείο τον Σερ Φράνσις Τζέικοψ, τον Τέο Νότεν και τον Τζον Καρ. Ε, παιδάκι μου, Να δώσουμε λοιπόν αμέσω το λόγο στο Σερ Francis Jacobs, ο οποίος είναι πρόεδρος του Missing Children Europe και ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, διότι μπορεί αργότερα να χρειαστεί να λείψω, έχουμε και άλλη ψηφοφορία. Παρακαλώ. Madam Chairman, it's a privilege for me to... Πρόεδρε, είναι χαρά μου να μπορώ να παραστώ σήμερα στη συνεδρίασή σας. Μετά από πολλά χρόνια ως γενικό εγγελέα στο δικαστήριο, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο που με απασχόλησε με πολλές τέτοιες επιθέσεις, έγινα πρόεδρος της, του Missing Children Europe, που είναι η οργάνωση που αφορά, ασχολείται με τα χαμένα, εξαφανισμένα παιδιά Έχουμε 24 ενώσει από τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν, από 16 κράτη-μέλη και από την Ελβετία. Έχουμε αρκετή εμπειρία με θέματα σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών και για παράδειγμα έχουμε λάβει ενεργό μέρος στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Συμμαχία που αναφέρθηκε από αρκετού ομιλητέ. Οι εθνικοί μας ε, οργανισμοί είναι, δραστηριοποιούνται στην πρώτη γραμμή και προσπαθούμε και εμείς να τους ενισχύσουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο ώστε να μπορούν να παρεμβαίνουν σε διασυνοριακά προβλήματα τα οποία αυξάνονται όσο μειώνονται τα σύνορα στην Ευρώπη και, που, και για να, εκπρο, ναι, μπορούν να εκπροσωπούν τα εθνικά του συμφέροντα ενώπιον του δικαστηρίου και της Κομισιόν. Έχουμε λοιπόν ασχοληθεί με πάρα πολλά τέτοια θέματα βέβαια παρόλο που δεν είμαστε απόλυτα, δεν έχουμε απόλυτα ομόφωνη φωνή, νομίζω ότι μπορούμε να μιλούμε με μια ευρωπαϊκή φωνή. Καλωσορίζουμε την προτινόμενη οδηγία που σκοπεύει να ε, καταστήσει την απόφαση πλαίσιο με την οποία, για την οποία είχαμε έρθει στη διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Καλωσορίζουμε τον νέο και σημαντικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη νέα διαδικασία λήψη αποφάσεων που ενισχύεται από την συνθήκη τη Λισαβόνα και καλωσορίζουμε αυτή την ευκαιρία για να μπορέσουμε και εμεί να το σχολιάσουμε. Στον χρόνο που έχω θα επικεντρωθώ σε μερικά σημεία. Βασικά θέματα νομικά, ε, αλλά και θέματα αρχής για να χρησιμοποιήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το χρόνο μου, δεν θα αναφέρω τα σημεία με τα οποία συμφωνούμε με τις υπόλοιπες μικρών, αλλά θα επικεντρωθώ στους τομείς με τους οποίους, ε, για τους οποίους ε, είτε δεν υπόθηκαν πολλά, είτε ε, ακόμη υπάρχουν συζητήσεις μεταξύ των μη κυβερνητικών οργανώσεων και για τις οποίες οι απόψεις διήστανται. Θα ξεκινήσω λέγοντας ε, ότι αναφέροντα αυτά που λέει και η Κομισιόν στο επεξηγηματικό μνημόνιο, ότι είναι σημαντικό και το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο ε, ως για αυτό το πολύ σημαντικό τομέα, ε, νομικό τομέα να έχουν υπόψη τους ότι τα συμφέροντα του παιδιού θα πρέπει να είναι ο βασικός τους στόχος σε οποιαδήποτε δράση αναλάβουν. Η αρχή αυτή αναφέρεται και στο άρθρο 24, παράγραφος 2 της Χάρτας των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης άρθρο 24, το άρθρο 24 λέει ότι τα παιδιά θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα σε τέτοια προστασία και φροντίδα, όπως, ε, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο, για όλες τις δράσεις που ασχολούνται με παιδιά και αναλαμβάνονται από ιδιωτικούς φορείς ή δημόσιες αρχές, το συμφέρον του παιδιού θα πρέπει να αποτελεί τη βασική πρόνοια. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σαφέστατα ε, ανέφερε τους, ποιοι είναι οι κανόνες ε, για την προστασία των παιδιών που δεν περιορίζονται μόνο σε μια ε, αρνητική αρχή της μη παρέμβασης αλλά περιλαμβάνει και μια θετική υποχρέωση να ποινικοποιούνται αδικήματα ενάντια στα παιδί ακόμη και προσπάθειες αδικημάτων. Η σεξουαλική κακοποίηση είναι ένα αναφυσβήτητο ε, αδίκημα με τεράστιες συνέπειες στα θύματα τους. Παιδιά ή άλλες ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες ε, δικαιούνται κρατική ε, προστασία μέσω με αποτελεσματικών αποτρεπτικών μέτρων και παρέμβασης. Μια τέτοια περίπτωση ήταν ε, η εναντίον της Φιλανδίας που έγινε το 2002 και μπορείτε να διαβάσετε την απόφαση ώστε να δείτε πώς ακριβώς το ε, δικαστήριο εξισορροπεί και την ελευθερία έκφρασης αλλά και την προστασία των δικαιώματων του παιδιού και πώς τα δικαιώματα του παιδιού αναγνωρίζονται ότι είναι ε, τα πιο σημαντικά. Τώρα, πάμε στην προτινόμενη οδηγία. Καταρχά, να πω ότι υποστηρίζουμε πλήρω την άποψη τη Κομισιόν ότι η οδηγία συνάδει με τι ε, αρχέ τη επικουρικότητα και τη αναλογικότητα. Σε ό,τι αφορά την επικουρικότητα, τα επιχειρήματα τη Κομισιόν στο επεξηματικό μνημόνιο ε, είναι απολύτω πιστικά. Όντω, σε ό,τι αφορά το ίντερνετ, ο τομέα όπου η επικουρικότητα ε, κατά περίπτωση έχει ανακληθεί θα ήταν δύσκολο να σκεφτούμε ε, ποια, πιο, ε, καλέ, πιο σωστές δράσεις σε, ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε ό,τι αφορά τώρα την αναλογικότητα, είναι προφανές ότι τα μέτρα που παρουσιάζονται στην οδηγία είναι απαραίτητα επίγοντα ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι και όντως εδώ δεν υπάρχει άλλο ένα επιχείρημα. Επίσης πρέπει να τονίσω την ανάγκη να εξασφαλίσουμε τη συνεκτικότητα με την, ε, με την, ε, με την, ε, συγγνώμη, με την σύμβαση του Λανσαρότε του Συμβουλίου. Είναι δεσμευτικό για κάποια κράτη-μέλη που πρέπει να αλλάξουν την νομοθεσία τους ώστε να συνάδουν με αυτό και να συμμορφωθούμε αυτό και κατά την άποψή μας θα ήταν καλό η οδηγία να είναι συνεπής και με την σύμβαση αυτή. Εκτός εάν υπάρχουν λόγοι όπου σε κάποια σημεία πρέπει να αναλυθούν διαφορετικέ δράσεις. Υπάρχουν πολλές, πολλά πλεονεκτήματα για μια τέτοια συνεκτικότητα, ώστε να μην υπάρχουν διαφορετικέ απόψει και μη συμβατέ απόψει για το ίδιο θέμα μεταξύ των κρατών μελών. Επίση, εισάγει ε, αβεβαιότητα σε, σε, στον τομέα του ποινικού δικαίου, όπου είναι ο τομέας όπου χρειάζεται απλότητα και σαφήνεια. Ε, δεν υπάρχουν δύο μέτρα και δύο σταθμά ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα δηλαδή για τα 27 μέλη της Ένωσης και ένα για τα υπόλοιπα 20 του Συμβουλίου της Ευρώπης και διευκολύνει την ε, υιοθέτηση της οδηγίας και την εφαρμογή της και πάνω απ' όλα υπάρχουν τομεί όπου η σύμβαση μπορεί να είναι προτιμότερη από το παρόν κείμενο τη οδηγία και κάποιε από τι τροπολογίε που έχουν ε, υποβληθεί. Υπάρχουν διάφορα θέματα ε, για την οδηγία όπου θεωρούμε ότι θα ήταν προτιμότερο να ακολουθήσουμε την ε, σύμβαση του λαθαρότε και όχι τις προτάσεις που έχουν γίνει μέσω της οδηγίας. Δεν υπάρχει τώρα χρόνος βέβαια να αναφέρω όλους αυτούς τους τομείς, αλλά θα ήθελα να τονίσω το θέμα αρχής ότι δηλαδή η συμφωνία, η συμμόρφωση με την ε, σύμβαση είναι ευκταίος στόχος. Αυτό φυσικά δεν υπονομεύει καθόλου την προστιθέμενη αξία της οδηγίας. Πολλά δε μάλλον όταν η οδηγία έχει το πλεονέκτημα ότι μέσω τη υιοθέτησή της από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι νομικός δεσμευτική από όλα τα κράτη-μέλη μπορεί να υπόκειται σε δράσεις εφαρμογή από την Κομισιόν σε περίπτωση που αυτό είναι απαραίτητο και θα υπόκειται σε ερμηνεία από το δικαστήριο ε, μετά από αναφορά των εθνικών δικαστηρίων ώστε να εξασφαλιστεί η σωστή και ομοιόμορφη ερμηνεία των διατάξεών της σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κάθε περίπτωση, όπως ε, ακούστηκε χτε από τους εκπροσώπους του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οδηγία δεν θα πρέπει να, ε, να υπολείπεται των, ε, των ορίων που υπάρχουν στο, στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης. Αυτό θα πρέπει να είναι το ελάχιστο και δεν θα πρέπει να υπαρξουν ρητρε ρήτρες opt-out. Θα πρέπει να υπάρχει ένα ενιαίο ομοιόμορφο πρότυπο. Επίσης, σύντομα να σχολιάσω κάποια ουσιώδη θέματα που θίγει η οδηγία. Καταρχήν, υπάρχει το θέμα της, των ελάχιστων ε, ε, ορίων, ε, των ελάχιστων ποινών ή των, ε, των ανώτερων ποινών. Ας πούμε, οι ανώτερες ποινές δεν θα πρέπει να είναι κάτω από 10 χρόνια κάθεξη. Γι' αυτό είναι σημαντικό για να δώσουμε ε, το σωστό μήνυμα, να, δώσουμε το, να δείξουμε το πόση σημασία δίνουμε σε αυτό το θέμα. Επίσης, θα πρέπει να ορίζονται ελάχιστες ποινές, που είναι τελείως διαφορετικό. Ας πούμε, η ποινή δεν θα πρέπει να είναι λιγότερη από δύο χρόνια. η ελάχιστη ποινή είναι άγνωστη στο ποινικό δίκαιο σε αρκετά κράτη-μέλη. Που, είναι, που θεωρούν σημαντικό το δικαστήριο να έχει την διακριτική ευχαίρεια να αποφασίζει και να προσαρμόζει τις ποινές σε όλες τις ε, περιπτώσεις που μπορεί να αξιολογήσει ένα τέτοιο δικαστήριο. Η ελάχιστη, μέγιστη ποινή δεν επηρεάζει αυτή τη διακριτική ευχαίρεια του δικαστηρίου. Αλλά ακόμη και για σεξουαλικά εγκλήματα που είναι ιδιαίτερω σοβαρά, η ελάχιστη ε, ποινή μπορεί να είναι λάθο σε κάποια περίπτωση. Μπορεί να υπάρχουν εξαιρετικέ περιπτώσει όπου οποιαδήποτε ε, κάθριξη δεν θα αποτελούσε τη σωστή ποινή και ίσω κάποια ε, φροντίδα ή κάποια θεραπεία εκτό φυλακή θα ήταν η ενδεδειγμένη συγκεκριμένη ποινή. Μπορεί να υπάρχουν επίση και θεμελιώδεις αντιρρήσει αρχή σε κάποια κρατημέλη για την εισαγωγή ελάχιστων ποινών. Δεύτερον, πιστεύουμε ότι θα ήταν σωστό να συμπεριλαμβάνονται διατάξει στην οδηγία που θα ε, διευρύνουν την, ε, το χρονικό περιθώριο ε, για σεξουαλικά εγκλήματα. Μια τέτοια διεύρυνση των χρονικών ορίων συνάδει και με τη σύμβαση του Λανθαρότε που καθορίζει ποια είναι η ε, που καθορίζει ότι η διοκτική αυτή διαδικασία μπορεί να τρέχει ε, μέχρι, για ικανοποιητικό χρόνο και μέχρι το παιδί να φτάσει σε περιγές περιπτώσεις και την ε, ηλικία ενηλικίωσης. Αν δηλαδή για, δεν, δεν μπορούν τα παιδιά να καταγγείλουν την, τα εγκλήματα που έχουν, των οποίων έχουν πέσει θύματα πριν φτάσουν στην ηλικία των 18. Το παιδί λοιπόν θα πρέπει να έχει τον απαραίτητο χρόνο, ώστε ακόμη και περιμένοντας για να ενηλικιωθεί, να μπορεί μετά να υποβάλει την καταγγελία του. Και να μπορούν αυτά τα εγκλήματα μετά να διώκονται. Το τελευταίο που θα ήθελα να αναφέρω είναι το ερώτημα της φραγής των ε, εικόνων ε, σεξουαλικής ε, παρενόχλησης. Ε, το μέτρο αυτό νομίζουμε ότι είναι ε, ένα ενδιάμεσο μέτρο ανάμεσα στην ε, διαγραφή και την αφαίρεση των εικόνων αυτών από το διαδίκτυο. Θέλω όμως να πω ότι ε, θεωρούμε ότι η φραγή είναι θεμελιώδες εργαλείο προστασίας για τα παιδιά θύματα. Ακούσαμε κάποιες αντιρρήσεις για, το, για τη φραγή. Χθες ακούσαμε ε, αντιρρήσεις λόγο της προστασίας των δεδομένων. Αλλά εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες και μέσα στο κείμενο της οδηγίας, το άρθρο 21 για παράδειγμα, παράγραφος 2, που ε, μπορούν να καθησυχάσουν αυτές τις ανησυχίες. Επίσης ακούσαμε για κάποιες αντιρρήσει που υπάρχουν λόγω ελευθερία ε, του λόγου και τη ενημέρωση. Αλλά θεωρούμε ότι είναι αδύνατο να λέμε ότι το να μπλοκάρει κανείς ε, εικόνες ε, σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, αυτές που εννοούμε εμείς εδώ, θα μπορούσε να θεωρηθεί περιορισμός της ελευθερίας της έκφρασης ή τη ενημέρωση. Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο ως επιχείρημα και βεβαίω δεν συνάδει καθόλου με τις αποφάσεις που έχει λάβει και το ε, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπινών Δικαιωμάτων για τέτοιες ε, υποθέσεις. Επίσης, δεν μπορούμε να δεχτούμε τα επιχειρήματα ότι αυτές οι εικόνες θα μπορούσαν ίσως ε, να... το μπλοκάρισμα τέτοιων ιστοσελίδων θα μπορούσε να οδηγήσει και στο μπλοκάρισμα ιστοσελίδων πειρατείας όταν υπάρχουν θέματα copyright, τζόγου κτλ αυτές οι περιπτώσεις θα πρέπει να, ε, να διερευνώνται η καθεμιά ξεχωριστά. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ε, δεν μπορούμε να μπλοκάρουμε το, τις ιστοσελίδες αυτές επειδή δεν θα μπορούμε να μπλοκάρουμε κάποιες άλλες ιστοσελίδες. Ε, οι ιστοσελίδες με εικόνες σεξουαλικής εκοπής είναι τελείως διαφορετικές. Mm-hmm. Οπότε θεωρώ ότι αυτά είναι θέματα αρχής. Υπάρχουν ε, και θέματα εξίσου σημαντικά, για τα οποία όμως δεν έχουμε χρόνο σήμερα να συζητήσουμε. Όπως ε, η ενηλικίωση που αναφέρθηκε ε, ήδη στην συζήτηση ή όταν θέλουμε να υπάρχει μία αναφορά στην ηλικία, την νόμιμη ηλικία για σεξουαλική δραστηριότητα. Επίσης θέλουμε να υπάρχουν διατάξεις για, την, ε, για το φιλτράρισμα των αιτήσεων εργασίας και, των, ε, και της ελεύθερης διακίνησης μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση τέτοιων ανθρώπων ε, που έχουν διαπράξει σεξουαλικά εγκλήματα. Οπότε αυτό χρειάζεται ένα ευρωπαϊκό σύστημα ελέγχου. Επίσης, κυρώσεις νομικών προσώπων, εταιριών, κατάσχεση του υλικού του εγκληματικού και επίση θα θέλαμε να τονίσουμε ότι πρέπει όλα αυτά να γίνονται άμεσα και οι έρευνε να διεξάγονται ε, γρήγορα. Αυτά είναι μερικά ε. θέματα για τα οποία θα θέλαμε να σα επιστήσουμε την προσοχή. Θεωρούμε ότι είναι πολύ χρήσιμη αυτή η ακρόαση. Επίση, ε, ελπίζουμε να έχουμε και άλλε ευκαιρίε να συμβάλλουμε στην δουλειά του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για αυτή την οδηγία. Και σα ευχαριστώ για την προσοχή σα. Oh, και εμεί σα ευχαριστούμε, κύριε Ιάκομψ. Και τώρα ο κύριος Τζον Κάρτ από την Ευρωπαϊκή Συμμαχία Μίκη μικρόν κατά της σεξουαλικής κακοποίησης παιδών. Ευχαριστώ την Επιτροπή σας για την τιμή που μου κάνει σήμερα να έχω την ευκαιρία να μιλήσω για αυτή τη σημαντική οδηγία. Θα, θα ακούσατε ότι εκπροσωπώ στην συμμαχία Μίκη Όμικρον κατά της κακοποίησης παιδών που αντιπροσωπεύει οργανώσεις από 20 περίπου χώρες και μέσα και έξω από την Ένωση. Πολλές από τις οργανώσεις αυτές παιδών ιδίως δε αυτές με τις οποίες έχω συνεργαστεί εγώ προσωπικά συνεργάζονται άμεσα με χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδων παιδών που έχουν τύχη σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή κακοποίησης σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή θυματοποίησης γενικότερα και το ίντερνετ συστηματικά έχει διευκολύνει τέτοιου είδους εκμετάλλευση και κακοποίηση. Πολλές από τις οργανώσεις με τις οποίες λοιπόν συνεργάζομαι ή τις οποίες εκπροσωπώ ασχολούνται και με την στενή παρακολούθηση των παιδιών αυτών, ψυχοθεραπευτικές μεθόδους και όλα τα άλλα που συζητούμε σήμερα. Ελπίζω λοιπόν στα σχόλια που θα σας κάνω να κατανοήσετε ότι δεν θέλω απλώς να μιλήσω ακαδημαϊκά ή αφηρημένα για, τις για τα σημαντικά θέματα αρχών που τίθενται εδώ, αλλά πρακτικά ολοκληρωτικά στην εμπειρία των παιδιών αυτών. Εμείς λοιπόν την οδηγία αυτή, το σχέδιο οδηγίας το θεωρούμε ως πολιτική πρόκληση, τι μας λέει, από πολιτικής απόψεως μας λέει ποιος θα δώσει φωνή στους αδύναμους και στα θύματα, στα παιδιά που υπέστησαν αυτά τα εγκλήματα όπως λέει το άρθρο 21. Η πολιτική είναι θέμα καθορισμού προτεραιοτήτων και εδώ τα πράγματα είναι καθαρά. Τι προτεραιότητα θα δώσει το Κοινοβούλιο στην προστασία των παιδών σε σύγκριση με άλλους στόχους. Και όπως και στη ζωή η πολιτική σημαίνει ότι θα υπάρχουν αντιτιθέμενοι στόχοι και προτεραιότητες. Το θέμα είναι να ληφθεί μια απόφαση ποια συμφέροντα, ποιες ομάδες θα προωθήσει κανείς περισσότερο από άλλα. Όλοι όσοι ασχολούνται βέβαια με το θέμα μας εκφράζουν τη λύπη τους και καταδικάζουν την ε, κακοποίηση και την εκμετάλλευση των παιδών, αλλά αυτά είναι λόγια. Είναι πολύ εύκολο να πει κανείς είμαι κατά, λυπούμε, γεια κλπ. Το θέμα όμως είναι τι γίνεται στην πράξη για να εμποδιστούν ή να καταργηθούν αυτές οι πρακτικές. Ας είμαστε λοιπόν σαφείς. Κανένα παιδί δεν δέχεται τέτοια εκμετάλλευση ή την ε, προβολή φωτογραφιών του με αυτόν τον τρόπο. Αν οι φωτογραφίες αυτές μπορούν να θεωρηθούν τουλάχιστον ως τρομερή παραβίαση του δικαιώματος του κάθε παιδιού στην ιδιωτική του ζωή, τότε οτιδήποτε βοηθάει την κυκλοφορία και διάδοση αυτών των εικόνων πρέπει να, να αντιμετωπιστεί. Για μας βέβαια και είναι γνωστό σε όλους μας η παρεμπόδιση, η καταστροφή αυτών των ιστοσελίδων είναι αυτό που θα προτιμούσαμε. Η απάλληψη όμως, η πλήρης απάλληψη όλων αυτών των πρακτικών δεν μπορεί να γίνει πρακτικά. Και όσο τα ψάχνουμε συνεχίζεται η διάδοση των εικόνων και η παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδών. Το δικαίωμά τους να αφαιρεθούν από το δημόσιο πεδίο αυτές οι εικόνες ταπείνωσης είναι βασικό δικαίωμα που μας δίνει ε, που μας κάνει να προτιμούμε την απάλληψη και όχι απλώς το μπλοκάρισμα. Το θέμα είναι πώς και τι θα γίνει στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή τέτοια απάλληψη. Και όσο δεν μπορεί να γίνει απάλληψη τότε θα προτιμούμε την, τόσο θα προτιμούμε τον μπλοκάρισμα. Πριν από μερικά χρόνια αυτή η τεχνολογία του μπλοκαρίσματος δεν ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη. Αλλά βλέπουμε ότι παραδείγματο χάρη η Deutsche Telekom χρησιμοποιεί κατάλογο μπλοκαρίσματος. Η Orange, η France Telecom επίσης. Η Telefonica στην Ισπανία και σε άλλες χώρες στον κόσμο χρησιμοποιεί τέτοιες καταλόγους, το Telecom Italia, το Google, τη Microsoft, η Τέλεια σονέρα στη Σκανδιναβία, η BT, η Vodafone, η Virgin. Τι θα τους πούμε τώρα, ότι επειδή δεν έχει αποδειχθεί η χρησιμότητα της τεχνολογίας αυτής πρέπει να τη σταματήσουν, όχι. Το μπλοκάρισμα και η φραγή εφαρμόζονται σε χώρες δημοκρατικές. Σουηδία, Δημοκρατία. Δανημαρκία, στην Ολλανδία και είναι παράλογο να λέει κανείς όπως υπονοούν ορισμένοι ότι αυτή η πρακτική οδηγεί σε παραβίαση δημοκρατικών δικαιωμάτων στην ελεύθερη έκφραση. Αυτά δεν ισχύουν. Είναι ένα μέσο που περιορίζεται αποκλειστικά στην παρεμπόδιση της διάδοσης παιδικής πορνογραφίας. Βέβαια, Σωστό είναι ότι υπάρχουν και άλλοι τρόποι, υπάρχουν τρόποι παράκαμψης μιας φραγής εμπλοκαρίσματος Πάντα μπορεί κανείς να βρει έναν τρόπο να δει αυτές τις εικόνες, αλλά εκατομμύρια ανθρώπων δεν το ξέρουν αυτό, δεν μπορούν να το κάνουν και άρα η φραγή δουλεύει. Επίσης ισχύει ότι υπάρχουν και άλλα μέρη του ίντερνετ όπως η τεχνολογία peer-to-peer peer to peer που μπορούν να παρακάμψουν τη φραγή και να χορηγήσουν μια κάλυψη χωρίς να φαίνεται και ποιος είναι ο χρήστης. Υπάρχουν όντως άλλα μέσα, αλλά αυτό δεν είναι λόγος να μην κάνουμε τίποτα εφόσον μπορεί να υπάρξει αποτέλεσμα. Κανείς δεν είπε ότι το μπλοκάρισμα πρέπει να επεκταθεί και στην τεχνολογία peer-to-peer. Το χρησιμοποιούμε ως μια σχετικά προσωρινή μέθοδο αλλά αποτελεσματική. Ορισμένοι ανησυχούν μήπως υπάρξει κατάχρηση του blocking σε χώρες ας πούμε όπου το πρόβλημα είναι ο τζόγος ή πνευματικά δικαιώματα στη μουσική και στο σινεμά. Εδώ θέλω να είμαι σαφής. Τι λέμε εδώ. ότι δεχόμαστε αυτή την τεχνολογία για τα δικαιώματα των παιδιών αλλά θέλουμε να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των τζογαδόρων ή ότι δεν θα εφαρμόσουμε αυτή την τεχνολογία για τα παιδιά χάρη στους τζογαδόρους εν ονόματι των τζογαδόρων. Οι εικόνες σεξουαλικής κατάχρησης ή εκμετάλλευσης παιδιών δεν είναι θέμα τζόγου, δεν είναι το ίδιο πράγμα. Δεν είναι κάτι που συζητιέται. Ούτε μπορούν να υπάρξουν ισοδυναμίες μεταξύ των παραβίαση των δικαιωμάτων των παιδιών και των δικαιωμάτων του Hollywood να αποφέρει κάποιο κέρδος. Δεν πρέπει να αφήσουμε τέτοιου είδους εξωτερικές σκέψεις όπως το πώς θα μπορούσε κανείς να καταχραστεί αυτή η τεχνολογία για άλλους τομείς. Τα παιδιά των οποίων οι εικόνες αναρτώνται στο ίντερνετ δεν έχουν καμία δυνατότητα προστασίας και δεν είναι δικαιολογία να πούμε ότι μπορεί η κυβέρνηση της Βόρειας Κορέας να καταχραστεί την τεχνολογία αυτή. Από τη δική μου περιορισμένη άποψη και από ό,τι γνωρίζω για τη Βόρεια Κορέα, νομίζω ότι δεν χρειάζεται τη βοήθεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για να καταχραστεί οτιδήποτε θέλει να καταχραστεί. Και δεν είναι το θέμα εδώ λοιπόν η τεχνολογία του μπλοκαρίσματος ή της φραγής. Τέλος είναι γελίο να λέμε ότι δεν πρέπει, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έναν καλό σκοπό η φραγή απλώς και μόνο γιατί ορισμένοι κακοί άνθρωποι τη χρησιμοποιούν για κακούς σκοπούς. Αν ακολουθήσουμε αυτό το επιχείρημα τότε και άλλα πράγματα, ορισμένα φάρμακα που χρησιμοποιούνται στην ιατρική, στα νοσοκομεία θα έπρεπε να απογορευτούν γιατί υπάρχουν οι τοξικομανείς. Τα όπλα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πολύ κακούς σκοπούς αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και κατά των αρουραίων. Δεν λέμε λοιπόν να απαγορευτούν τα όπλα επειδή ορισμένοι κακοί άνθρωποι τα χρησιμοποιούν για κακούς σκοπούς. Νομίζω ότι αυτό γίνεται εσκεμμένα για να συγχυστούν τα πράγματα. Επομένως δεν είναι δικαιολογία αυτό το επιχείρημα. Εφόσον ο σκοπός μας είναι κάλλιστος. Καταλήγω λοιπόν ξαναλέγοντας ότι πρόκειται για πολιτικό θέμα και επιλογής του Κοινοβουλίου. Ποιον θα επιλέξει. Ελπίζω να επιλέξει να προστατέψει τα θύματα, τα παιδιά δηλαδή των οποίων οι εικόνες αναρτώνται παράνομα στο Ιντερνετ. Ευχαριστούμε πολύ. Και τώρα ο τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Τέο Νότ, από το ECPAT International, End Child Prostitution, Pornography and Trafficking. Ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε το λόγο και τη δυνατότητα να σας απευθύνω κάποια πράγματα. Βέβαια δεν έχω και τίποτα να προσθέσω. Οι προλαλήσαντες έχουν πει σχεδόν τα πάντα για το blocking να πω ότι υποστηρίζω, όπως είπαν και οι συνάδελφοι, το blocking. Να πω ότι απογοητεύομαι που βλέπω τόσο λίγο ευρωβουλευτές στην αίθουσα. Τι σημαίνει το πρόβλημα δεν θεωρείται κάτι σημαντικό. Uh, I know that there were some... Ξέρω ότι υπήρξαν προβλήματα με την κίνηση σήμερα, αλλά εγώ ήμουνα στις 8 η ώρα εδώ. 8. Δυσκολεύτηκα να ξυπνήσω, αλλά ήρθα. Να πω λοιπόν ότι ο οργανισμός μας είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός που προσπαθεί να σταματήσει την παιδική πορνογραφία, την πορνογραφία και την εκμετάλλευση των παιδιών ε, για σεξουαλικούς σκοπούς καθώς και του σεξουαλικό κορισμό, τουρισμό. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι τα παιδιά απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους χωρίς να υπάρχει καμία εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση. Έχουμε οργανισμούς και δίκτυα σε πάνω από 75 χώρες παγκοσμίω και έχουμε ενεργά μέλη στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε 15 χώρες. Θα μιλήσω σήμερα για το πρόβλημα του παιδικού σεξουαλικού τουρισμού. Είναι η εκμετάλλευση παιδιών ε, και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά έχουμε εκμετάλλευση και σε τρίτε χώρε. Πολίτε δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση που εκμεταλλεύονται και κακοποιούν παιδιά σεξουαλικώ στο εξωτερικό. Σεξουαλικό τουρισμό έχουμε σε ανθρώπους που ταξιδεύουν από τη μία χώρα στην άλλη και ε, εκμεταλλεύονται σεξουαλικώς παιδιά. Ορισμένες φορές γίνεται διαφοροποίηση μεταξύ σεξουαλικού τουρισμού και ε, παιδικής ε, πορνείας. Δυστυχώς το φαινόμενο μπορεί να εμφανιστεί σε πάρα πολλές χώρες και σε πολλές περιπτώσεις έχουμε και διασύνδεση με την εμπορία. Ε, υπάρχει εμπορία παιδιών σε τουριστικούς προορισμούς διότι εκεί πληρώνονται περισσότερο οι σεξουαλικές υπηρεσίες που προσφέρονται ακριβώς επειδή βρίσκονται σε τουριστικό προορισμό ε, σε ένα θέρετρο διακοπών ή ακόμα και σε ένα ε, χώρο επαγγελματικών ε, δραστηριοτήτων, αλλά Πολλές φορές δεν σημαίνει απαραίτητο ότι ταξιδεύουν εκεί για να βρουν τα παιδιά. Πολλές φορές μπορούν να τα βρουν και μέσω διαδικτύου ή μπορούν να εκμεταλλευτούν τα παιδιά ακόμα και στο ίδιο τους το σπίτι οι εικόνες σεξουαλικής κακοποίησης αυξάνονται και μάλιστα σε αντίστοιχο ρυθμό με το σεξουαλικό τουρισμό. Τα παιδιά μπορεί να είναι θύματα δηλεμπορίας ε, απλώς και μόνο για να έχουμε περισσότερο πορνογραφικό υλικό. Η παιδική πορνογραφία λοιπόν συνδέεται και μεταξύ, ε, με το σεξουαλικό τουρισμό και το εμπόριο παιδιών. Είναι πολλά υποσχόμενο το θέμα της αντιμετώπισης του σεξουαλικού τουρισμού, διότι πολλές χώρες έχουν νομοθεσία. Αλλά ε, η αστυνομία μπορεί να δράσει μόνο αν δεν υπάρξουν ε, καταγγελίες. Δυστυχώς όμως οι χώρες στις οποίες υπάρχει ο σεξουαλικός τουρισμός ε, δεν είναι εξοικειωμένοι με το ε, με το σύστημα του σεξουαλικού τουρισμού. Διότι τι μπορεί να κάνει κάποιο όταν βλέπει ένα 50χρονο, πούμε, να κάθεται με μια 15χρονη κοπέλα που μοιάζει με 30χρονη ε, και ε, υπάρχει κάποια σεξουαλική δραστηριότητα. Σε κάποιε περιπτώσει δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Η συνεργασία λοιπόν σε τοπικό, εθνικό και διεθνέ επίπεδο είναι απαραίτητη για να μπορέσουν να συλληφθούν οι άνθρωποι αυτοί και να καταδικαστούν. Ορισμένες φορές δεν υπάρχουν δυνατότητες, δεν υπάρχει συνεργασία με κάποιες χώρες, δεν υπάρχει εναρμόνιση της νομοθεσίας και ε, υπάρχει πρόβλημα και με την ηλικία συγκατάθεσης. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Η συνεργασία μεταξύ αστυνομικών δυνάμεων και μη κυβερνητικών οργανώσεων ε, θεωρείται απαραίτητη η συνθήκη για να μπορέσουμε να ε, καταλήξουμε σε καταδίκη αυτών των ανθρώπων. Οι αστυνομικέ δυνάμεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ε, διασυνδέσεις που έχουν με τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις για να επιταχυνθούν διαδικασίες. Παραδείγματο χάρη, ο κύριος Τ. κάτοικος του Ηνωμένου Βασιλείου ήταν μάρτυρας μιας σεξουαλικής κακοποίησης ε, στην Καλκούτα το 2006. Ο κύριος Τι το κατήγγειλε στην τοπική αστυνομία και στο αυστριακό ε, προξενείο, αλλά δεν αναλύθη καμία δράση. Μετά από μήνες, ο κύριος Τι, ο οποίος ήταν αστυχαίο ήρθε σε επαφή με την ε, ΕΚΠΑΤ, του Ηνωμένου Βασιλείου και η ΕΚΠΑΤ του Ηνωμένου Βασιλείου και η ΕΚΠΑΤ της Αυστρίας ε, εργάστηκαν και κατάφεραν να ξεκινήσει μια διαδικασία ανάκρισης και το 2007 μετά από κάποια χρόνια καταδικάστηκε ε, ο δράστης ε, στην Αυστρία ε, σε καταδίκη χωρίς δυνατότητα αναστολής. Θεωρούμε λοιπόν ότι η συνεργασία είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και η οδηγία επίσης ε, ε θεωρείται σημαντικό βήμα για την καταπολέμηση του σεξουαλικού τουρισμού και θα θέλαμε να υπάρξει και μια εναρμόνιση με τη σύμβαση του Λανθαρότε. Θεωρούμε όμω ότι και κάποια πράγματα θα πρέπει να προχωρήσουν λίγο περαιτέρω. Στο άρθρο 2, για παράδειγμα, στου ορισμού, θα θέλαμε να οριστεί ο σεξουαλικό τουρισμό ως σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών από άτομο ή άτομα από το συνήθες τους περιβάλλον σε ένα προορισμό όπου υπάρχει σεξουαλική επαφή με τα παιδιά. Στο άρθρο 3, στα αδικήματα που σχετίζονται με τη σεξουαλική κακοποίηση, θα θέλαμε η ηλικία συγκατάθεσης ε, να αφαιρεθεί διότι ορισμένες φορές ε, ε, δεν θα έχουμε εναρμονισμένη προστασία των παιδιών σε όλη την Ευρώπη και μπορεί να έχουμε και κακοποίηση σε χώρες στις οποίες οι ηλικία συγκατάθεση είναι χαμηλότερη από τη χώρα σας. Το άρθρο που αναφέρεται στη σεξουαλική εκμετάλλευση. να τιμωρείται ο πελάτης που ε, χρησιμοποιεί σεξουαλικές υπηρεσίες παιδιών, ε, διότι υπάρχει μεγάλη προετοιμασία για την αγορά σεξουαλικών υπηρεσιών. Άρθρο 6 που αναφέρεται στην εκμετάλλευση των παιδιών για σεξουαλικούς σκοπούς. Εδώ θα πρέπει να υπάρχει αναφορά, ε, να μην υπάρχει συγγνώμη αναφορά στην ηλικία συγκατάθεσης βάσης διεθνούς δικαίου και η προστασία θα πρέπει να ισχύει για όλα τα παιδιά και τα παιδιά είναι όλα τα άτομα κάτω των 18 ετών στο άρθρο 7 ε, παραπλάνηση και ε, άλλες διευθετήσεις. Ε, δεν ε, έχουμε ταξίδια μόνο για να διαπράψει κάποιος τα δικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 2 6. Έχουμε και άλλα δικήματα. Κυρώσεις σε νομικά πρόσωπα. Ε, προσωρινή ή μόνιμη πάυση λειτουργίας ε, καταστάσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη διάπραξη του αδικήματος θα πρέπει να προσθεθούν εδώ. Στο άρθρο 14, έρευνα και ε, καταγγελίες και δίωξη, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ειδικέ ευαίσθητε ε, μονάδες ε, στην αστυνομία, να υπάρχει κατάλληλη επιμόρφωση στο δικαστικό και αστυνομικό προσωπικό, όπως δηλώνεται και στην, ε, στην αντίστοιχη δήλωση. Όσον αφορά τώρα τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τους επαγγελματίες, θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικές απαιτήσεις και θα πρέπει να ισχύει αυτό για λόγους ομοιομορφίας στην όλη Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης θα θέλαμε να αποσυρθεί το άρθρο 16.3 που δίνει τη δυνατότητα του opt-out, διότι αυτό μπορεί να παρακολύσει την προστασία ε, σε κάποιες περιπτώσεις. Τώρα, στο άρθρο 10 ε, τις απαγορεύσεις που προκύπτουν από τις καταδίκες. Τα μέτρα αυτά θα πρέπει να ισχύουν για όλες τις δραστηριότητες ε, που αφορούν ε, συχνή επαφή με τα παιδιά. Εάν ε, υπάρχει δράση ο οποίο καταδικάζεται για τα αδικήματα που αναφέρονται στα άρθρα 3 έως 7 θα πρέπει να υπάρχουν ε, εγγραφές σε μητρώα ε, δραστών σεξουαλικών αδικημάτων. Κάποια επαγγέλματα, όπως παραδείγματο χάρη οδηγή, ταξί, γονεί, θύματα τα οποία συλλαμβάνονται για μικροαδικήματα και άλλες αστυνομικέ δυνάμει πρέπει να χρησιμοποιούνται διότι είναι πολύ δύσκολο να συλλέξουμε στοιχεία όταν έχουμε αρκετές χώρες που εμπλέκονται στη διαδικασία. η χήμη κυβερνητικών οργανώσεων, ε, κάποια προσοχή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικά για να καταλήξουμε σε καταδίκη. Πολλές φορές η σύλληψη και η καταδίκη είναι συνεργασία σε πολλά επίπεδα ε, και εθνικά αλλά και διεθνώς. Πολλές φορές κάποιοι διαφεύγουν της χώρας ή αποφεύγουν την κράτηση ή καταφέρνουν ε, το θύμα να αποσύρει την καταγγελία του. Και αν κάποιος βγει με αναστολή ε, και με εγγύηση μπορεί να καταφέρει να διαφύγει. Ε, οι παραβάτες λοιπόν που συλλαμβάνονται και βγαίνουν με εγγύηση θα πρέπει ε, να αποφεύγονται, διότι θα πρέπει να υπάρχει επίσης και κατάλληλη μέρημνα ώστε να επιστρέφουν τελικά στην ε, συνηθισμένη τους ζωή χωρίς να διαπράττουν αδικήματα. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μπορεί να διαδραματίσει πολύ σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να διασφαλίσει ότι η οδηγία αυτή θα έχει τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Σα ευχαριστούμε που μα δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσουμε και να συνδράμουμε στο θέμα αυτό. Σα ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. μην κρίνετε την απουσία των Ευρωβουλευτών σήμερα γιατί δυστυχώς σήμερα έχουμε ταυτόχρονα πολλές ψυχοφθορίες στο Κοινοβούλιο και γι' αυτό λείπουν. Τώρα θα δώσω το λόγο στον κύριο Μπρόντσο. το πρόεδρε Ο κύριος Σέλστρομ μας είπε 1852 άτομα έχουν ταυτιστεί από εικόνες και είπε ότι αυτός ο αριθμός είναι μικρός. Α, έχει φύγει βλέπω, τέλος πάντων. Πόσο μικρός θα ήθελα να ρωτήσω και γιατί. Ο δε κύριος Ρόμπινς χρησιμοποίησε τον όρο URL, νομίζω ότι πρέπει να ομολογήσω δεν ξέρω τι σημαίνει. 98,6% είπατε χρηστών ευρείας πρόσβασης, ταχείας πρόσβασης ε, σωστό ήταν, ε, συνεργάζονται για την ε, παρεμπόδιση τέτοιων ιστοσελίδων. Άρα το υπόλοιπο 4% δεν το πράττει. Δεν συνεργάζεται με προμηθευτές που καταπολεμούν. Αυτό το κάνουν επίτηδες, δηλαδή επιλέγουν προμηθευτάς που να μην συνεργάζονται ή απλώς, ή απλώς τους επιλέγουν αθώα. Και άρα ερωτώ ποιοι είναι αυτοί οι προμηθευτέ που δεν συνεργάζονται. Είναι συνένοχοι των παρονόμων αυτών δραστηριοτήτων ή είναι απλώς απρόσεκτοι και ο κύριος Μακνάμι μίλησε για τις φραγές και την παρεμπόδιση πρόσβασης ε, στο σελίδες που δείχνουν τέτοιο περιεχόμενο. Για, τους, για τα μονοπόλια τζόγου γνωρίζει τίποτα, έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ για πολιτικούς στόχους οι φραγές για να μην μπορούν οι πολίτες να έχουν πρόσβαση σε μια πολιτική ιστοσελίδα. Αν ναι, τότε εγώ θα ήμουν κατά. Από την άλλη όμως πρέπει να συμφωνήσω ότι το γεγονός ότι υπάρχει κατάχρηση σε μερικούς τομείς δεν είναι λόγος για να μην χρησιμοποιηθεί η τεχνολογία αυτή σε αυτόν τον τομέα. Είπε βέβαια κάποιος και κάτι άλλο. Depacket είπε κάποιος. Depacket inspection. Και πριν από μια εβδομάδα συνάντησα τον όρο αυτόν, από ό,τι κατάλαβα, εννοεί ότι πρόκειται για αυτόματη εξέταση της ιστοσελίδας στην οποία έχει κάποιος πρόσβαση για να δει αν έχει τέτοιο περιεχόμενο. Αλλά εντάξει καλό είναι αυτό εφόσον βέβαια αυτή η επιτήρηση δεν χρησιμοποιείται και για άλλους σκοπούς. Αν δηλαδή για να δουν αν η κυβέρνηση εγκρίνει ή όχι τις ιστοσελίδες. Α, ναι, και κάτι άλλο δεν ναι. ναι, ναι κύριος Νότον είπε, μίλησε για τη σύνδεση πορνείας και παιδοπορνογραφίας. Σε μερικές πόλεις και κομοπόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο υπάρχουν νεαρές κοπέλες, έφηβες, που τους ναρκώνουν αφού τους ε, πουν διάφορα ρομαντικά και καταλήγουν στην πορνεία. Σε μερικές πόλεις είναι αυτό γνωστό, σε άλλες όχι. Όταν οι καταχρήσεις αυτές προέρχονται από ευαίσθητες περιοχές, καμιά φορά η αστυνομία διστάζει να παρέμβει, καθώς και τα μέσα μαγικής ενημέρωσης να αναφέρουν. Τελεία. Α, εγώ θα αρχίσω εγώ. Το URL είναι ένας όρος που εννοεί τη διεύθυνση μιας ηλεκτρονικής σελίδας. Είναι ένας τεχνικός όρος, μια τεχνική έκφραση. Εννοεί διευθύνση σελίδων, αυτό θα πει URL. Με περιεχόμενο εικόνες, γράμματα, αριθμούς. Αυτό εννοούμε URL, διεύθυνση. Λοιπόν, για να είμαστε σαφείς τώρα για το 98,6%. Το 98,6% των Άγγλων προμηθευτών έχει αξιολογηθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και είδε διαπίστωσε ότι η καταναλωτές που τους χρησιμοποιούν καλύπτονται από εταιρείε που βρίσκονται στον κατάλογο, που χρησιμοποιούν τον κατάλογό μας. Άρα, όντως, φαινομενικά τουλάχιστον, οι προμηθευτέ αυτοί έχουν ελεγχθεί. Βέβαια δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα γιατί το υπόλοιπο 1,4% συμπεριλαμβάνει μεταπολιτές υπηρεσιών του κυρίου προμηθευτού. Και δεν έχουμε φτάσει μέχρι τέτοια λεπτομέρεια ελέγχου για να δούμε δηλαδή αν και αυτό το 1,4% είναι επιλήπουσιμο. Αλλά το 98,6% είναι πολύ καλός αριθμός εφόσον μάλιστα πρόκειται για εθελοντική κάλυψη. Υπάρχει και μία ιστοσελίδα που δείχνει τα ονόματα των προμηθευτών αυτών για να μπορούν οι καταναλωτές και καταναλώτριες, οι χρήστες και οι χρήστριες να τα βλέπουν. Δεν ξέρετε όμως αν αυτό το 1,4% είναι συνένοχοι σε τέτοιες παρανομίες ή να απλώς απρόσεκτοι. Όχι, δεν θα έλεγα ότι είναι συνένοχη στη διάδοση τέτοιων φωτογραφιών ή πορνογραφιών. Αλλά θα το δούμε στο μέλλον για να φτάσουμε το 100%. Για να δούμε δηλαδή γιατί αυτοί δεν καλύπτονται. Με συγχωρείτε που επανέρχομαι, ε, γιατί δεν υπάρχουν και άλλοι εξάλλου, αλλά αυτοί που χρησιμοποιούν αυτό το 1,6%, 1,4%. Χρησιμοποιούν αυτούς τους προμηθευτές γιατί έτσι έτυχε ή το επιλέγουν επίτηδες. Ε, κοιτάξτε, αυτό συζητιέται, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν ξέρω αν όντως επίτηδες επιλέγουν αυτούς τους προμηθευτές που δεν υπάρχουν στον κατάλογό μας. Ναι, αλλά αν υπάρχει αυτή η υποψία, τότε θα μπορούσατε να στοχεύσετε αυτούς τους προμηθευτάς. Ναι, αν ισχύει αυτό, ναι. Ο κύριος Γαόλ. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν ποιος είναι σε αυτό το 1,4% και αν επιλέγουν επίτηδες αυτούς τους προμηθευτές για να έχουν πρόσβαση σε σελίδες πορνο, παιδοπορνογραφίας. Αλλά πριν από μερικά χρόνια είχε διαπιστωθεί ότι οι εικόνες αυτές παιδοπορνογραφίας είναι στα news groups που είναι ένα ειδικό ιδιαίτερο μέρος τμήμα του ίντερνετ και πριν αναλάβει ο Πίτερ τη διεύθυνση της οργάνωσης του είχα ασχοληθεί και εγώ και το Internet Watch είχε αρχίσει να μπλοκάρει την πρόσβαση σε αυτά τα news groups που έχουν τέτοιες φωτογραφίες και η αστυνομία μας είπε ότι μερικοί υποπτευόταν ότι όντως επέλεγαν προμηθευτές που δεν κάνανε τη φραγή αυτή δεν είναι, δεν είναι δηλαδή αβάσιμη υπόθεση να πει κανείς ότι μερικοί επιλέγουν επίτηδες αυτούς τους προμηθευτές που δεν χρησιμοποιούν τη φραγή και ότι οι, χρήστε χρήστες αυτών των προμηθευτών το κάνουν επίτηδες. Κύριε Μακνάμι μήπως θέλετε κι εσείς να πείτε τίποτα. χρονομέτρησα για να δω πόσος χρόνος χρειαζόταν για να αλλάξω τις ρυθμίσεις μου στο ίντερνετ και μόνο 27 δευτερόλεπτα χρειάστηκαν για να αποφράξω επιλήψιμο περιεχόμενο. Νομίζω λοιπόν ότι δεν είναι μεγάλο εμπόδιο. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα ιστοσελίδων που έχουν φραχθεί κατά λάθο, που δεν έχουν επιλήψιμο περιεχόμενο. Δύο όμως παραδείγματα φραγών που ποτέ δεν περιείχαν τέτοιο περιεχόμενο υπάρχουν και παραδείγματος χάρη η μόνη ιστοσελίδα που έχει φραχθεί στο Βέλγιο λέγεται σταματήστε την περδοπορνογραφία αυτή η σελίδα έχει φραχθεί εδώ και πολύ καιρό γιατί παραβίαζε του νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων ορισμένων κρατουμένων αλλά αποφράχθηκε την περασμένη εβδομάδα και μετά επαναφράχθηκε και μετά επαναποφράχθηκε χωρίς να έχει αλλάξει το περιεχόμενό της. Φαίνεται δηλαδή ότι πότε είναι νόμιμο, πότε παράνομο. Να, ένα παράδειγμα. Belgian blocking page is really worth the visit. Ναι, λοιπόν, η ιστοσελίδα αυτή είναι σε τέσσερις γλώσσες και λέει, έχει μια προειδοποίηση που λέει εδώ προσπαθείτε να μπείτε σε μια σελίδα που παραβιάζει το βελγική, τη βελγική νομοθεσία. Αν είστε ο ιδιοκτήτης της ιστοσελίδας παρακαλώ στείλτε μας ένα τηλομοιότυπο. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τρομερά ενδιαφέρον. Ο ιδιοκτήτης λοιπόν της ιστοσελίδας ο ίδιος δεν έχει λόγο να δει ποτέ αυτή την προειδοποίηση αφού δεν είναι στη χώρα Εδώ τώρα μιλάμε για εγκλήματα σοβαρά, για παρανομίες που ε, ιστοσελίδων που εδρεύουν σε άλλες χώρες και τι μας λένε εδώ. Ας γνωρίζουν οι παρανομούντες ότι παρανομούν. Και αν θέλουν να μας στείλουν ένα φάξ. Αυτό μας φαίνεται πολύ μυστήριος τρόπος αντιμετώπισης του προβλήματος. Και το άλλο παράδειγμα είναι φιλανδική ιστοσελίδα που λέγεται κάτι σαν παιδοπορνογραφία.com και μεταξύ άλλων επικρίνει και τους φραγμούς, τις φραγές. Να, αυτά είναι τα δύο παραδείγματα. Αυτά. Α, όχι αυτά, όχι αυτά υπάρχει και η διάδοση σε άλλους κυβερνοχώρους. Αν η Κομισιόν θεωρεί ότι είναι αρκετά σημαντικό το θέμα της φραγής για να ώστε να ζητάει και υπόσχεση ότι δεν θα υπάρξει επέκταση της τεχνολογίας αυτής σε άλλους τομείς ενώ ταυτόχρονα χρηματοδοτεί προγράμματα φραγής τότε αυτό πρέπει να το ξέρει το Κοινοβούλιο. Αν παίρνει πρωτοβουλία στο Συμβούλιο μπλοκαρίσματος άλλων περιεχομένων εκτός της περδοπορνογραφίας, τότε και εσείς πρέπει να το ξέρετε αυτό για να μπορέσετε να, κάνετε, να βγάλετε την απόφασή σας. Δεν πρόκειται λοιπόν για εξισορρόπηση αλλά για το ότι η Κομισιόν λέει κάτι που θεωρεί σωστό και ταυτόχρονα λέει ότι δεν ισχύει. Ευχαριστώ πολύ και τώρα η κυρία Ζήπελ. Ευχαριστώ. Δυστυχώς δεν άκουσα όλες τις ε, παρουσιάσεις, αλλά θα ήθελα να επανέλθω σε αυτό που ακούστηκε σήμερα το πρωί από μία εκπρόσωπο η οποία είπε ότι πρέπει να έχουμε μεγαλύτερη ευαισθησία, πρέπει να βρούμε νέα μέτρα, αλλά η όλη συζήτηση για αυτό το πολύ ευαίσθητο θέμα δεν θα πρέπει να καταλήξει σε ιστερία. Και αυτή είναι μια εμπειρία που συχνά την βλέπουμε σε τέτοιες περιπτώσεις κακοποίησης, όπου καταλήγουμε να, να ποινικοποιούμε ανθρώπους που δεν έχουν τελικά καμία σχέση με το αντικείμενο και αυτό κάνει τη δουλειά μας πολύ δυσκολότερη. Νομίζω ότι με την οδηγία αυτή έχουμε το εξή πρόβλημα. Έχουμε τον τίτλο της οδηγίας, ο οποίος ε, δεικνύει μια πολύ ευρεία προσέγγιση. Μιλούμε για πρόληψη, μιλούμε για αντιμετώπιση σεξουαλικής κακοποίησης, μιλούμε για εκμετάλλευση, που επίσης ένα άλλο, είναι μια άλλη πτυχή, μιλούμε για τον πραγματικό κόσμο και την κακοποίηση σε αυτόν τον πραγματικό κόσμο. Μιλούμε για την αντιμετώπιση της ε, ε, ζήτησης τέτοιων ε, ιστοσελίδων στον ψηφιακό κόσμο, στο ίντερνετ. Τις τελευταίες εβδομάδες η συζήτηση έχει επικεντρωθεί κυρίως στο ίντερνετ και, και το τι κάνουμε με το διαγραφή ή φραγή των ιστοσελίδων. Εγώ πρέπει να ε, πω ότι η τεχνική αυτή συζήτηση με την, ε, ε, με την όλη διαδικασία φραγής ή διαγραφής είναι περισσότερο περίπλοκη παρά χρήσιμη. Δεν ξέρω αν πρέπει να επικεντρωθούμε στο αν είναι σωστό να γίνεται διαγραφή ή φραγή, αλλά αν με αυτή την οδηγία μπορούμε να δημιουργήσουμε μία ε, δικαιολογία ώστε να φράσονται στο μέλλον και άλλοι ε, τομεί και άλλε τοσελίδες που εκπίπτουν του πεδίου εφαρμογή αυτή τη οδηγία. Εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Νομίζω ότι πρέπει να δώσει η Κομισιόν ένα σαφέ μήνυμα. Εάν θέλει να ε, φράξει, τι ακριβώς θέλει να φράξει και αν μπορεί αυτό να γίνει με την αυτόματα. Δηλαδή, ο αυτοματισμό υπάρχει. Να το χρησιμοποιήσουμε σήμερα για να μπλοκάρουμε μια ιστοσελίδα πορνογραφικού υλικού, αύριο για να μπλοκάρουμε κάτι άλλο. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε αυτό, γιατί πραγματικά έχουν ενταθεί πολύ οι απόψει και στη συζήτηση που γίνεται. Και ένα άλλο σημαντικό, χτες ακούστηκε το θέμα της πρόληψης. Μιλούμε για διαγραφή αλλά και για ποινικά μέτρα. Αυτά είναι κάποιες πτυχές αυτού του, αυτού του θέματος. Έχουμε συζητήσει πάρα πολύ για το θέμα της πρόληψης, ότι πρέπει όντως να συμπληρωθεί η πτυχή αυτή, αλλά ένα πολύ σημαντικό σημείο και νομίζω ότι εκεί πρέπει να κάνουμε ακόμη περισσότερες συζητήσεις και με τα κράτη-μέλη και το κάναμε και χτες και το κάναμε και ακούσαμε και σήμερα α, τους να το λένε, το επειδή ακριβώς δεν μιλούμε μόνο για την ε, ε, πραγματική ε, κακοποίηση γιατί μιλούμε κυρίως για την κακοποίηση στο ίντερνετ που σχετίζεται και με την εμπορία προσώπων κτλ. Εάν θέλουμε να, να προχωρήσουμε και να μειώσουμε τις, τους αριθμούς των θυμάτων κακοποίησης στο ίντερνετ ή στον πραγματικό κόσμο. Χρειαζόμαστε όμως έμπειρο ε, προσωπικό, χρειαζόμαστε ε, διοκτικές αρχές και αυτό δεν μπορεί να ρυθμιστεί μόνο μέσω της οδηγίας. Τα κράτη-μέλη είναι αυτά που έχουν την ε, υποχρέωση να έχουν ένα αξιόπιστο, μια αξιόπιστη προσφορά σε όλους αυτούς τους φορείς που χρειάζονται για την αντιμετώπιση των θυμάτων των υποθέσεων κακοποίησης. Συγγνώμη. Και ένα πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Μιλήσαμε και για το ποινικό δίκαιο, για την όξυνση των ποινών. Ε, θα ήθελα να μου πείτε εάν όσοι είσαστε σήμερα εδώ στο Προεδρείο μπορείτε να μου πείτε από την εμπειρία σας εάν έχετε αριθμούς, αν έχετε ε, συγκεκριμένα στοιχεία για το αν όντω αξίζει τον κόπο να οξυνθούν οι, υψηλέ ε, ψηλές γιατί ίσω αυτέ οι ποινέ, αν είναι πολύ υψηλέ, να καταστήσουν πιο εύκολο το να δολοφονηθεί το παιδί για να εξαφανιστεί ας πούμε ο μάρτυρα που θα μπορούσε να τον στείλει τον ε, δράστη αυτό στη φυλακή. Οπότε μήπω έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία για να δούμε ότι όντω με την όξυνση των ποινών μειώθηκαν τα θύματα κακοποίηση. Ευχαριστώ πολύ. Μήπω θέλετε να προσθέσετε κάτι, ο κύριο Μακναμή, ο Σερ Τζέικοπς. Παρακαλώ. Ο κύριος Νότεν, χωρίς μικρόφωνο. Ξέρω ότι στις κάτω χώρες υπάρχει ποινή για κατοχή ε, παιδικής πορνογραφίας και η διανομή παιδικής πορνογραφίας ε, έχει αυξηθεί γιατί είναι σχεδόν ε, αυξήθηκε μάλλον συγγνώμη, η ποινή γιατί υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν και άλλα ερευνητικά μέσα. Αν θέλει κάποιος για παράδειγμα να εξετάσει περιβάλλον peer-to-peer -peer, πρέπει να υπάρχει ψηλότερη ποινή. Τουλάχιστον αυτό βάσει Ολλανδικής νομοθεσίας. Εμείς έχουμε μια αντίστοιχη κατάσταση στο Ηνωμένο Βασίλειο. Για να μπορέσει κάποιος ε, να ενταχθεί σε προγράμματα θεραπείας ε, ατόμων που έχουν διακράξει σεξουαλικά δικήματα, ε, πρέπει να έχεις λάβει συγκεκριμένη ποινή. Δεν ξέρω αν υπάρχει άμεση ε, σχέση με το επίπεδο της, ε, του αδικήματος. Από νομικής πλευράς δεν υπάρχει τίποτα. Επειδή ο κύριος Σάλστρομ είναι και αυτός ακόμα εδώ, μήπως θέλετε να προσθέσετε κάτι για την πείρα σας ε, στη Σουηδία, για στοιχεία, για φραγές. Έχετε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία. Όχι, δεν έχω. Ανάλογη συζήτηση γίνεται και στη Σουηδία όμως ε, για τις ε, δυνατότητες έρευνας. Δυστυχώς για να μπορέσεις να ερευνήσεις κάποια πράγματα περαιτέρω πρέπει να έχουμε ε, περισσότερα χρόνια ποινής. Υπάρχουν ερωτήσεις από πλευράς μελών ή δεν ξέρω αν θέλετε να ακούσουμε και κάποιους άλλους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λαντσμπέργκης λέγομαι, από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Κατά λάθο παρατηρητής εδώ, θα ήθελα να κάνω μία μικρή παρατήρηση, αν μου επιτρέπετε. Μπορώ? Παρακαλώ. Η παρατήρησή μου είναι η εξή. Παιδική πορνογραφία σε ιστοσελίδε. Υπάρχουν ε, πραγματικά ε, πάροχοι, σερβερς, χρήστες. Ε, Η άποψή μου είναι ότι είτε πρόκειται για ερασιτέχνες είτε για επαγγελματίε. Business makers δεν θα έπρεπε καν να αποκαλούνται επισήμως ε, server providers. Πώς μπορούν να σταματήσουν αυτές οι υπηρεσίες. Εύκολο. Ίσως είναι νομοθετικό το πρόβλημα. Αλλά όσοι διανέμουν τέτοιο υλικό δεν θα πρέπει να θεωρούνται ε, ως provider ε, συγκεκριμένου σερβερ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Πολ Ντουράντ. από του Ιρλανδούς Service Providers ε, και διαχειρίζομαι επίσης και έναν οργανισμό ο οποίος ασχολείται με δημόσιες διαμαρτυρίες για ε, δημόσιο περιεχόμενο στο διαδίκτυο. Ε, σήμερα όμως εκπροσωπώ την Euroest, του Ευρωπαϊκή Οργάνωση Internet Service Providers που εκπροσωπεί αρκετές οργανώσεις παγκοσμίων. Καταρχάς να πω ότι χαιρετίζουμε την οδηγία, διότι περιλαμβάνει κατά την άποψή μας πολλά άρθρα που αφορούν τη σεξουαλική εκμετάλλευση στον πραγματικό κόσμο. Εμείς δεν είμαστε εμπειρογνώμονες στο τομέα, αλλά ο πραγματικός κόσμος είναι η πηγή των εικόνων που συζητούνται τόσο πολύ και στη συνέχεια διανέμονται στο διαδίκτυο. Ε, από αυτή την άποψη ε, είμαστε οι εμπειρογνώμονες για το διαδίκτυο. Να πω κατηγορηματικά σε όλους ότι τα μέλη της Γιουρέσπα σε καμία περίπτωση δεν θέλουν να κυκλοφορεί αυτό το υλικό στα δίκτυά μας. Και μάλιστα εμείς έχουμε πάρα πολύ πρακτική πείρα ε, σε στενή συνεργασία με την αστυνομία για να προσπαθήσουμε να διαγράψουμε το υλικό αυτό από τα δίκτυά μας. ως τεχνικοί εμπειρογνώμονες, εμείς θεωρούμε ότι τα μόνα μέτρα τα οποία ε, αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά την κυκλοφορία τέτοιου υλικού είναι να αφαιρεθεί στην πηγή του το συντομότερο δυνατόν. Οποιοδήποτε άλλο μέτρο είναι καλοπιστική φύσεω για διάφορου λόγου που ακούσατε σήμερα, διότι αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα, μετακινούνται πολύ γρήγορα εικόνε. Δεν είναι αποτελεσματικά λοιπόν αυτά τα μέτρα. Το πρόβλημα επίση που υπάρχει με το μπλοκάρισμα είναι ότι η παράνομη πηγή μένει ανέπαφη ε, και αυτοί που θέλουν πρόσβαση και έχουν πρόσβαση στο υλικό αυτό μπορούν να το μετακινήσουν πάρα πολύ γρήγορα και να το ε, αντιγράψουν σε άλλη στο σελίδα. Το υλικό λοιπόν εξακολουθεί να υπάρχει και οι δράστες ε, ουσιαστικά τελικά μένουν ατιμόρυτοι, ενώ τα παιδιά τα οποία έχουν να υπάρξει αντικείμενο κακοποίηση ε, είναι έρμεο αυτών των ανθρώπων και οι εικόνε του κυκλοφορούν ακόμα στο διαδίκτυο. Εμεί λοιπόν θα θέλαμε η οδηγία αυτή να ενισχυθεί σε κάποιου τομεί κυρίως σε θέματα διαδικτύου και θεωρούμε ότι το βασικό θέμα εδώ είναι ότι θα πρέπει να επικεντρωθούμε ε, στην ανάπτυξη ενός σαφούς νομικού και δικαστικού πλαισίου για να κατεβαίνουν πάρα πολύ γρήγορα αυτές οι εικόνες από το διαδίκτυο και να συλλαμβάνονται οι δράστες από τις αποδείξεις που αφήνουν στο διαδίκτυο. Να μην ε, μπλεχτούμε σε πάρα πολύ τεχνικές λεπτομέρειες δηλαδή, αλλά να επικεντρωθούμε στο πιο συνολικό θέμα για ποιο λόγο ακούσαμε κάποιους να λένε ότι το να κατεβάσουμε μια ιστοσελίδα δεν λειτουργεί πάρα πολύ γρήγορα. Πού είναι ο ανακριτής να πει ότι ορίστε πού υπάρχουν προβλήματα, γιατί δεν κατεβαίνει γρήγορα το ιστοσελίδα. Θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το πιο αποτελεσματικό μέτρο πρέπει να εστιάσουμε στα αποτελεσματικά μέτρα και να μην σπαταλούμε χρόνο και χρήμα σε πράγματα τα οποία δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Ολοκληρώνοντας λοιπόν να πω ότι εμείς ως Γιουρίσπα θα θέλαμε να ζητήσουμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Κοινοβούλιο να έχει πάντα κατά νου ότι κάθε ευρώ που σπαταλάτε σε καλοπιστική μορφή μέτρα θα έπρεπε να χρησιμοποιείται για να χρησιμοποιήσουμε την πιο αποτελεσματική μέθοδο και να προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε την αποτελεσματική μέθοδο ώστε τα παιδιά να μην ε, αποτελούν περαιτέρω αντικείμενο εκμετάλλευση. Και αυτό είναι να βρίσκουμε το υλικό στην πηγή του, να κατεβαίνει και να διαγράφεται και η αστυνομία να βάζει τους δράστες εκεί που ανήκουν, πίσω από τα δυσφυλακή στα σίδερα. Ε, Um, Πρόεδρε, ευχαριστώ που μας καλέσατε σήμερα στην ακρόασή σας. Για εμάς που δουλεύουμε στον τομέα της προστασίας του παιδιού είναι πραγματικά πολύ σημαντική αυτή η ακρόαση. Εγώ δεν ξέρω πολλά από κομπιούτερ, η αλήθεια είναι, αλλά αυτή που Αυτά που ακούστηκαν ε, με ανησύχησαν λίγο, όπως τα είπε ο κύριος Μακναμία, α πούμε. Ξέρει πώς λειτουργεί η τεχνολογία ο ναι. ίδιος. Αλλά κάποιοι από τους, αλλά και κάποιοι από τους ε, προηγούμενους το ρώτησαν. Τι θα γίνει όμως αν δεν περάσει η οδηγία. Μπορεί εντάξει να μην είναι τέλεια, να έχει κάποια τεχνικά προβλήματα, αλλά αν ε, μπλοκαριστεί είτε λόγω τεχνικής, τεχνολογίας είτε λόγω προστασίας δεδομένων, τι θα γίνει. Ξέρω τι λέει ο κύριος Κάρ, κατανοώ ποια είναι η θέση του και τον υποστηρίζω 100% αλλά μετά από μια σημαντικά τεχνική ακρόαση, εμείς που απλώς νοιαζόμαστε για τα παιδιά, ποια εναλλακτική θα έχουμε. Δεν ξέρω αν μπορούν να μαντέψουν, να διακινδυνεύσουν ε, να μαντέψουν οι παριστάμενοι. Προφανώς όλες οι ε, οργανώσεις συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε κάτι και το χρειαζόμαστε άμεσα. Αλλά τι θα είναι αυτό. Πριν ε, δώσω το λόγο στους ομιλητές, Πρέπει να ζητήσω για άλλη μια φορά συγγνώμη, αλλά δυστυχώ υπήρχαν οι ψηφοφορίε ε, και γι' αυτό δεν ήμουν εδώ. Να ε, καθησυχάσω τη μέρη μπανότη. Θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μα για να εκρίνουμε την οδηγία εγκαίρω και ο λόγο για τον οποίο έχουμε αυτέ τι μέρε συζήτηση, οι οποίε κατά την άποψή μα θα πρέπει να συνεχιστούν, είναι να συνεργαστούμε όλοι από κοινού, ώστε να έχουμε ένα κείμενο που ε, μα αφορά όλου, το οποίο θα είναι χρήσιμο και αποτελεσματικό. Αυτή είναι η προτεραιότητα του Κοινοβουλίου και θα συνεργαστούμε με όλου όσου χρειάζεται, ώστε να επιτύχουμε το κατάλληλο αποτέλεσμα προ το συμφέρον των ανηλίκων κυρίω, προ το συμφέρον των θυμάτων, αλλά και για να προλάβουμε ε, καταστάσεις στις οποίες θα υπάρχουν θύματα. Ποιος θέλει το λόγο? Um, <clears throat> Δεν νομίζω ότι έχω τόσες τεχνικές γνώσεις όσες ε, μου αποδίδεται, αλλά όλοι τον ίδιο στόχο έχουμε. Κάτι πρέπει να υπάρξει ώστε να προχωρήσουμε μπροστά γρήγορα. Ακούσαμε και τις ε, συζητήσεις ε, που έχουν γίνει και από την Επιτροπή Εκπαίδευσης και Πολιτισμού. Έχει γίνει λοιπόν πολύ καλή δουλειά για να υπάρξει συμβιβασμός και φαντάζομαι, ελπίζω ότι το Κοινοβούλιο θα ε, καταλήξει σε κάτι αρκετά χρήσιμο. Δεν θέλω να επαναλάβω αυτό που λέει ο κύριο Ντουράν, αλλά χρειαζόμαστε όντως μια σωστή αξιολόγηση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε στο ίντερνετ. Πολλές φορές ε, οι πολίτες καταγγέλουν σε ευρωπαϊκές γραμμές βοήθειας τι παράνομε ιστοσελίδε, περνάνε από μια λυσίδα επικοινωνία και σε, κάποιο, σε κάποιες περιπτώσεις ε, προκύπτει κυρίως από τη ΣΥΠΑ οι ιστοσελίδες αυτές να παραμένουν online. Δεν έχει γίνει όμως έρευνα για να δούμε πού βρίσκονται τα προβλήματα. Προσπαθούμε να βρούμε λύση χωρίς να ξέρουμε ποιο είναι το πρόβλημα που θέλουμε να λύσουμε. Η λύση του εισφραγής, όπως είπε και ο κύριος Ρόμπιν χτες, βασίζεται στο πώς είχαν τα πράγματα πριν από τέσσερα χρόνια, όπου όλα τα domain names ξεκινούσαν από ένα σημείο. Και αυτό δεν συμβαίνει πια. Ή συμβαίνει όλο και λιγότερο. Οπότε λύνουμε ένα πρόβλημα που ουσιαστικά έχει τροποποιηθεί και δεν βασίζουμε τη λύση μας σε έρευνες που να, ασχολούνται με το πώς έχει η κατάσταση τώρα. Εγώ συνεργάζομαι συχνά και πολύ καλά με τους παριστάμενους εδώ στο πάνελ και πρέπει, συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να υπάρχει μια περιοδική ε, αναφορά και προς τα κρατημέλη και προς την Κομισιόν ώστε να ξέρουν όλοι τι ακριβώς γίνεται σε διεθνές επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Γιατί προς το παρόν πολλές ε, χώρες ε, δεν παρουσιάζουν τίποτα αλλά Μόνο αν επικεντρωθούμε στο να έχουμε αυτά αποτελέσματα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Να δούμε δηλαδή ποιες είναι, ποια είναι τα αποδεκτικά στοιχεία, να δούμε πώς μπορούμε όντως να πιάσουμε τους ανθρώπους αυτούς και να τους στείλουμε στη δικαιοσύνη, όχι να κάνουμε ασκήσεις επί χάρτου. Ευχαριστώ. Έχουμε μία ακόμα παρέμβαση από τον κύριο Μπάλς. Πολλά ακούστηκαν για τα θύματα. Εγώ εκπροσωπώ την οργάνωση Μόργους και ονομαζόμαστε η φωνή των θυμάτων. Για μας το πρόβλημα είναι ότι συνεχώς μιλάνε υπέρ ημών, αλλά δεν μας δίνουν το λόγο. Εμείς θέλουμε να αυτοεκπροσωπηθούμε. Είναι η Μόρκους μια γερμανική οργάνωση που δεν τίθεται υπέρ της φραγής, γιατί δεν έχει εμποδίσει την εκμετάλλευση. Έχει γίνει πολλής λόγος για την αποτελεσματικότητα της απάλληψης Δεν καταλαβαίνω γιατί τίθενται προβλήματα για την απάλληψη. Εγώ ξέρω τι συμβαίνει και τα χειρότερα ακόμη και δεν καταλαβαίνω γιατί περιορίζεστε στην κατάρτιση ενός καταλόγου αντί να απαλήφετε. Εξάλλου στον κατάλογο αυτό των χειροτέρων περιπτώσεων και μια άλλη γερμανική οργάνωση που είναι κατά της φραγής εξέτασε τον, κατάλογο, τον δανέζικο κατάλογο είχε 160 περίπου στο σελίδες πολλές από τις οποίες δεν είχαν καμία σχέση με παιδοπορνογραφία εξάλλου πολλές από αυτές τις ιστοσελίδες δεν λειτουργούσαν πια Τρεις από αυτές τις ιστοσελίδες μπόρεσαν να απολυφθούν μέσα σε 30 λεπτά. Μία δε Ολλανδική που ζήτησε να φραχθεί μεταφέρθηκε στην Ινδία. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν ποιο πρόβλημα έχει η αστυνομία να αντιδράσει εγκαίρως. Η απάλληψη των σελίδων είναι κάτι εύκολο. Εξάλλου κάτι ανάλογο είπε και ο κύριος Μακναμή. Πρέπει να δούμε ποιο είναι πρώτα το πρόβλημα και μόνο τότε μπορούμε να μιλήσουμε για λύση του. Εγώ δεν νομίζω ότι η φραγή είναι λύση. Είναι δικαιολογία για να μην αντιδράσει κανείς και εγώ δεν θέλω να υπάρχουν εδώ τέτοιες δικαιολογίες. Τα παραδείγματα από τη Δανία και τη Σουηδία το δείχνουν η φραγή δεν εμποδίζει, ενώ η απάλληψη μπορεί να γίνει σε μισή ώρα μέσα. Υπάρχουν σελίδες που είναι στον κατάλογο 1,5 χρόνο και συνεχίζουν να αναρτούν το περιεχόμενό, τους, το περιεχόμενό τους. Γιατί δεν κάνει τίποτα η ασουτινομία. Ήθελα να κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπόλτ. Τον γνωρίζω και τον ευχαριστώ πολύ και για τη δέσμευσή του, αλλά και γιατί έχει το θάρρος να πολεμάει από πλευρά θυμάτων γιατί έχει υπάρξει και ο ίδιος θύμα. Θεωρώ όμως ότι από τη συζήτηση που είχαμε εδώ αυτές τις δύο μέρες Κανένας δεν θεωρεί ότι το blocking είναι η μία και μόνη λύση. Όλοι μας είπαν ότι ο βασικός στόχος είναι να διαγράψουμε το περιεχόμενο και να μην διατίθεται. Δηλαδή, να πάμε στην πηγή και να αφαιρέσουμε αυτό το περιεχόμενο. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι εφικτό κάτι τέτοιο, διότι μπορούμε να βρούμε την πηγή, γιατί οι αρχές συνεργάζονται γέρος. Σε κάποιες όμως περιπτώσεις δεν είναι δυνατόν, διότι ε, μπορεί να πρόκειται για εγκληματική οργάνωση, μπορεί να μην είναι γνωστή η πηγή, μπορεί να μην υπάρχει συνεργασία με την χώρα προέλευσης. Είναι δυστυχώς μια σειρά από γραφειοκρατικά προβλήματα αυτά. Και εδώ μας είπαν όλοι ότι ούτως ή άλλως πρέπει όμως να προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο να το αφαιρέσουμε. Αλλά στο ενδιάμεσο διάστημα μέχρι να φτάσουμε στην πηγή θα πρέπει να μπλοκάρουμε με κάποιο τρόπο την ιστοσελίδα. Με κάποιο τρόπο να διαγράψουμε ακόμα και αν αυτό γίνεται για προσωρινούς λόγους. Το δεύτερο στοιχείο που κατεμένει σημαντικό είναι αυτό που ακούσαμε να λέγεται ότι ακόμα και όταν ε, δηλαδή αφαιρείται το περιεχόμενο, έχουμε φτάσει στην πηγή και έχουμε αφαιρέσει το περιεχόμενο, επειδή ακριβώς είναι τόσο εύκολο να το αντιγράψουμε, μπορεί να ξαναεμφανιστεί μετά από λίγες μέρες, μετά από λίγες ώρες, ακόμα και μετά από κάποιους μήνες. Δηλαδή, το μπλοκάρισμα ούτως ή άλλως δεν είναι το μέσο ή μάλλον το μόνο μέσο είναι ένα συμπληρωματικό εργαλείο για να επιτύχουμε τον αρχικό μας στόχο. Αυτό για να σας ρωτήσω τι. Εσείς είστε ούτως ή άλλως ε, κατά του blocking, ακόμα και αν πρόκειται για το προκαταρκτικό στάδιο πριν από τη διαγραφή. Δηλαδή εσείς προτιμάτε, ακόμα και αν χρειάζεται ένας μήνας για να διαγράψουμε το περιεχόμενο, για αυτό το μήνα να αφήσουμε την, το περιεχόμενο στο διαδίκτυο και να μην παρέμβουμε με κανένα τρόπο. Mm. Αυτό θα θέλατε. So, first, I would like to... Καταρχάς, να ρωτήσω γιατί σας παίρνει ένα μήνα. Αν έχουμε για phishing για χρήματα από τράπεζες, αυτές ε, οι σελίδες κατεβαίνουν σε 4 με 8 ώρες παγκοσμίως. Γιατί χρειάζεται ένας μήνας για να κατέβει μία εικόνα ενός παιδιού. Ε, κατ' εμέ πρόκειται για αποτυχία διεθνούς συνεργασίας, αποτυχία διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας. Η Interpol κάνει blocking σε 188 χώρες. Έχει 118 μέλη που κάνουν blocking. Ε, πρώτα αφαιρούμε και μετά κοιτάμε τι περισσεύει. Οποιαδήποτε χώρα η οποία έχει ε, οποιαδήποτε αστυνομική δομή είναι μέλος της Ιντερπολ. Γιατί πρέπει να διορθώσουμε, ε, να επισκευάσουμε ένα κουβά και γιατί δεν πετάμε κατευθείαν τον κουβά. Ε, έχουμε σελίδες οι οποίες βρίσκονται παγκοσμίω σε όλο τον κόσμο. Το blocking δεν είναι ένα μέτρο που ζητούν τα θύματα. Τα θύματα ε, γνωρίζουν ότι το blocking δεν είναι η λύση, διότι το πρόβλημα δεν είναι ότι οι, σελίδες, οι εικόνες βρίσκονται σε μια συγκεκριμένη σελίδα, αλλά το πρόβλημα είναι η ίδια ύπαρξη των εικόνων. Και ξέρουμε όλοι ότι υπάρχουν οι σελίδες ότι μπορούν να βρεθούν οπουδήποτε, ακόμα και σε έντυπη μορφή. Κάποιος μπορεί να σας στείλει σπίτι με το ταχυδρομείο. Ε, η πρόσβαση είναι το πρόβλημα και το blocking ε, δεν ε, είναι λύση. Μπορώ να σας το πούνε τα περισσότερα θύματα. Μπορώ να σας το πω από την πείρα μας, αλλά τα περισσότερα θύματα είναι κατά του blocking. Μπορεί να σας εκπλήσει, αλλά είναι, είμαστε κατά του blocking και ως ενδιάμεση λύση, διότι θα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που λειτουργεί το διαδίκτυο. Θα πρέπει να αλλάξει η υποδομή του διαδικτύου και υπάρχει μια κεντρική αρχή που μπορεί να ελέγξει το περιεχόμενο. Εγώ είμαι από τη Γερμανία. Η Γερμανία Γερμανία βίωσε δύο δικτατορίες ή μάλλον ε, περίπου δικτατορίες ε, ε, σε 50 χρόνια. Εγώ είμαι από την πρώην Ανατολική Γερμανία, ζούσα σε σοσιαλιστική χώρα, σε μια χώρα όπου υπήρχε έλεγχος πληροφοριών. Κανένας δεν θέλει να έχει τέτοια εξουσία στο διαδίκτυο. Αυτό είναι το διαδίκτυο. Πρόκειται για ένα μεγάλο μέσο εκδημοκρατισμού και αυτό είναι το πρόβλημα. Το εσείς αυτή τη στιγμή παραβιάζετε το ίντερνετ, παραβιάζετε το πιο όμορφο πράγμα που έχουμε. Το διαδίκτυο είναι ένας τρόπος να επικοινωνούν οι άνθρωποι και ολοκληρώνοντας να πω υπάρχουν καλές και κακές πτυχές αλλά δεν θα πρέπει να ε, δημιουργήσετε προβλήματα στο ίντερνετ διότι οι κατα... ε, κακοποιήσεις συμβαίνουν στην πραγματική ζωή. Και παρά το γεγονός ότι εμείς είμαστε θύματα κακοποίησης ε, παιδιών έχουμε δικαιώματα και τα παιδιά έχουν δικαιώματα και εσείς ε, παραβιάζετε το ίντερνετ ε, το δικό μας. Το stopkinderporn.com είναι η μόνη στο σελίδα που δεν βρίσκεται στη σελίδα μπλοκαρίσματος. Πότε μπαίνει, πότε βγαίνει. Μίλησα στον ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι από τις κάτω χώρες και ε, ορισμένες φορές ε, μιλάει με τα θύματα. Μπορεί να ε, υπερβάλλει στον τρόπο με τον οποίο καταπολεμά ε, την κακοποίηση γιατί βάζει τους δράστες στο διαδίκτυο, αλλά στο Βέλγιο δεν κάνουν μπλοκάρισμα σε υλικό και νομίζω ότι ε, βλέπετε γιατί είναι τόσο επικίνδυνο το μπλοκι. Δεν υπάρχει νομική διαδικασία. Υπάρχει το μπλοκάρισμα στο Βέλγιο και ο συγκεκριμένος άνθρωπος από, την Ολλανδία δεν μπορεί να καταπολεμήσει αυτή την... Ε, ε ε, τη λίστα, λέει δεν υπάρχει νομοθεσία και ο Υπουργό λέει ότι α, να σας μπλοκάρουμε στο μέλλον. Μπορεί να είναι κακό, μπορεί να είναι το ίδιο πρόβλημα που είχαμε και στη Φιλανδία. Ο Μάρτιν Νίκη πήγε στην αστυνομία και είπε εάν μπλοκάρετε την ε, ε, σελίδα μου ουσιαστικά ε, κυκλοφορούν πληροφορίες στο ίντερνετ και τον έχουν στον κατάλογο και δεν μπορούν να παρέμβει. Δεν έχει κανένα μέσο να παρέμβει. Και να πω και κάτι για το Μόγκους. Ε, εμείς θεωρούμε ότι το άρθρο 6 είναι πάρα πολύ κακό. Δεν θα σταματήσει η κακοποίηση των παιδιών. Θα έχετε ένα άρθρο το οποίο θα τρομάξει τους ανθρώπους που εργάζονται και έχουν συναντήσεις με τα παιδιά. Ε, γιατί τα παιδιά δεν θα έχουν σε ποιον να στραφούν. Εάν θέλει κάποιο να μιλήσει εμπιστευτικά για τη σεξουαλική κατακοποίηση, θα πρέπει να κάνει μια συνέντευξη ένα προ ένα. Δεν θα την κάνει δημόσια. Εάν ε, κάποιο θέλει να κάνει συζήτηση με τα παιδιά είτε στο διαδίκτυο είτε εκτό διαδικτύου, τότε αφαιρείται ουσιαστικά από τα παιδιά την προστασία που χρειάζονται. Σα ευχαριστώ πολύ. Thank Σας ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να, να μιλήσω επιτέλους για το θέμα του κλίματος στην κοινωνία όπου γίνονται αυτές οι παραβιάσεις. Αυτό το αρνητικό κλίμα που προωθούν τα μέσα με αυτή την μη ρεαλιστική παρουσίαση της πραγματικότητας για ανθρώπους δηλαδή που τόσο εύκολα φτάνουν σε σεξουαλικές συναντήσεις. Έχουν πολλούς σεξουαλικούς εταίρους. Αυτό που λέμε δηλαδή προμισκούιτι μεταξύ γυναικών και ανδρών και που είναι άνθρωποι που δεν έχουν καν καρδιά. Δεν προσκολώνται σε κανέναν. Αυτό δεν το ανέφερε καμία παρουσίαση. Το θέμα λοιπόν είναι αν κάποιες συμπεριφορές είναι αποδεκτές για οποιονδήποτε άνω των 18 τότε πολλοί θα αναρωτηθούν γιατί να μην είναι αποδεκτές και από τους 17 ή και τους 16 και 15 Αυτό το κλίμα είναι που αφορά τις σεξουαλικές επαφές που σε πολλές περιπτώσεις θεμελιώνει αυτές τις παραβιάσεις. Ευχαριστώ. Έχουμε μία ακόμα παρέμβαση από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ο κύριος Αλόνσο Ριάρτε. Ε, πρέπει να σεβαστούμε και λίγο το χρονοδιάγραμμα. Στις 12.30 θα πρέπει να ολοκληρώσουμε την ακρόαση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ήδη ακούστηκε η φωνή της Κομισιόν, απλώς δύο πραγματάκια θα ήθελα να θέξω. Καταρχήν και αυτό το κίνδυνο στο ίντερνετ που αναφέρεται. Ακούστηκαν κάποια αρθεντικά στοιχεία από την Eurostat για το ποσοστό όσων χρησιμοποιούν το ίντερνετ κατά μέσο όρο κάθε μέρα. Αν πάρουμε έξι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ε, χρησιμοποιούν εντατικά το ίντερνετ, Σουηδία, Ολλανδία, Δανία, Λουξεμβούργο, Φιλανδία και ε, Ηνωμένο Βασίλειο. Σε αυτές τις έξι χώρες Υπάρχει μεγάλη χρήση ίντερνετ. Ε, Τέσσερι ναι. χώρε έχουν σύστημα φραγή. Οπότε προφανώ δεν πλήττεται η εμπιστοσύνη του, ανθρώπου, του κόσμου στο ίντερνετ και ο κατάλογο αυτό ε, των χωρών που έχουν ε, συστήματα φραγή για την παιδική πορνογραφία δεν είναι χώρα καταλόγων που καταπατούν την ελευθερία τη έκφραση, κάθε άλλο παρά. Απλώ ήθελα να σα το υπενθυμίσω γιατί. η οδηγία δεν ε, προσπαθεί να καλύψει μια κατάσταση όπου ε, λειτουργούν τα πάντα τέλεια. Δεν είναι οδηγία για έναν ιδεατό κόσμο, είναι οδηγία για μια ε, κοινωνία όπως είναι τώρα. Και όπως είναι ο κόσμος τώρα, αν κάνουμε κάτι για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση όπως έχει. Ή απλώς αν ευχόμαστε ότι η κατάσταση θα ήταν διαφορετική, να ήταν καλύτερα. Ε, οι ευχές όμως δεν βοηθούν τα παιδιά. Υπάρχουν άλλε παρεμβάσει. Νομίζω πως όχι. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους τους προσκεκλημένους μας και να ανανεώσω την πρόσκληση ε, που έκανα σε όλους να στείλετε στη γραμματεία της Επιτροπής μας και τις ε, παρεμβάσεις ε, όλων των προσκεκλημένων μας. αλλά και οποιαδήποτε περαιτέρω συνεισφορά ό,τι έχετε ευχαρίστηση προκειμένου να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε το κείμενο της οδηγίας να συμφωνήσω απολύτως με τα τελευταία λόγια του Αλόλ Σοριάρτε εμείς εδώ βρισκόμαστε για να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Προφανώς αυτή η οδηγία θα επικαιροποιηθεί, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συνεργαστούν και με τη σειρά τους να αναλάβουν και αυτά δεσμεύσεις. Καταλαβαίνουμε τον κόσμο του διαδικτύου, τον κόσμο της τεχνολογίας ε, και ε, ξέρουμε ότι είναι ένας κόσμος ο οποίος εξελίσσεται συνεχώς, αλλά θα πρέπει να γίνει κάτι, είναι απαραίτητο και αυτή είναι η δέσμευση που έχουμε αναλάβει εμείς από πλευρά Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Σίγουρα δεν θα κάνουμε την τέλεια οδηγία, αλλά θα προσφέρουμε χρήσιμα εργαλεία για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε το φαινόμενο της online κακοποίησης και γενικότερα της εκμετάλλευσης των ανηλίκων. Ευχαριστώ πολύ.